Good afternoon, everyone. I'm very pleased to welcome you all. Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε την ακρόασή μας για τον αντίκτυπο της ε, αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ε, στην, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους εμπειρογνώμενες που είναι εδώ μαζί μας σήμερα για τη σημαντική αυτή ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Στις 29 ε, Μαρτίου, τα μεσάνυχτα ε, του 2019, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσει μια τρίτη χώρα. Αυτό δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, κυρίως ως προς τον αντίκτυπο της αποχώρησής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκφύσεως είναι διασυνοριακά και το αποτέλεσμα φυσικά είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές μας, την βιωσιμότητα των πολιτικών μας ή ε, την ποιότητα και τις προδιαγραφές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι βέβαιη ότι ε, ίδιες είναι και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε οργανώσει τη σημερινή ακρόαση για να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε ε, αυτόν τον αντίκτυπο της του Brexit ε, στις ε, πολιτικές ε, που είναι της αρμοδιότητός μας θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες ε, που θα λάβουμε σήμερα στους διαπραγματευτές μας, ε, ώστε αυτά τα ζητήματα να αντανακλώνται ε, σωστά στις διαπραγματεύσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο αρνητικός αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα το πώς θα λάβει η χώρα η σημερινή ακρόαση, 10 λεπτά θα έχει κάθε ομιλητής για να κάνει την παρουσίασή του και κάθε δύο παρουσιάσεις θα έχουμε ερωταποκρίσεις στις οποίες μπορούν οι βουλευτές να λάβουν το λόγο. Εγώ περιμένω με πολύ χαρά τη σημερινή συζήτηση και χωρίς να καθυστερήσω άλλο να δώσω το λόγο στον πρώτο μας προσκεκλημένο που είναι ο κύριος ε, Πέτερ Γιόρτ Κάλσεν, ο εκτελεστικός ε, ε, αναπληρωτής διευθυντής της Europarla Foods. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να σας ε, παρουσιάσω ε, την ε, άποψή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε ένα συνεταιρισμό, σε Arla Foods, ε, εγώ είμαι επικεφαλής της ε, στην ε, Ευρώπη και πιο πριν ήμουν επικεφαλής της Arla Foods στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε γνωρίζω και ε, τις δύο πλευρές και ξέρω και τους καταναλωτές των δύο πλευρών. Για την Arla Foods λοιπόν, το να υπάρχει ένα, μια ασφαλής, ε, ένας ασφαλής βιώσιμος γαλακτοκομικός τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το υψηλό επίπεδο της, ε, των τροφίμων, της ε, ασφάλειας των τροφίμων ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό από τότε που αρχίσαμε το 1880 με, μια, με ένα πάρα πολύ μικρό ε, συνεταιρισμό. Επειδή η ασφάλεια των τροφίμων ήταν τμήμα του ταξιδιού από την αρχή, το Brexit ε, ήρθε κατά κάποιο τρόπο ως έκπληξη ε, τον Ιούνιο του 2016 για μας. Ως Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός εμείς βασιζόμαστε σε αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Δεν αποτελεί μυστικό ότι θα, θα προτιμούσαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εργαστούμε σκληρά για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή μελλοντική σχέση σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου με σεβασμό της ακαιρεότητα Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ενιαία αγορά. Θα ήθελα σύντομα να σα παρουσιάσω την, το συνεταιρισμό Arla Foods και τη σημασία του Brexit ε, Φυσικά θα αναφερθώ μετά στο ενδεχόμενο αντίκτυπο της ε, αποχώρησης ε, του ε, Ηνωμένου Βασιλείου στον συνεταιρισμό μας. Η Arla Foods είναι μια γαλακτοκομική εταιρεία με ιδιοκτήτες αγρότες, 11.200 αγρότες από 7 κράτη-μέλη της Ένωσης, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σουηδία, Δανία και Μπενελούξ. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την υψηλότερη δυνατή αξία για το γάλα των γεωργών μας. Προσπαθούμε να πληρώσουμε την υψηλότερη τιμή καθημερινά. Το κέρδος μοιράζεται μεταξύ των γεωργών, μεταξύ όλων των 7 χωρών. 170 ε, μέλη έχει το Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπροσώπων, ε, εκπροσωπώντα τους 11.200 γεωργού ε, που και λαμβάνουν όλε τι όλες τις βασικές αποφάσεις. Έχουμε κατά κάποιο τρόπο το δικό μας μικρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντό του συνεταιρισμού. Οι γεωργοί μα ε, παρέχουν 14 δισεκατομμύρια κιλά γάλακτο, η τέταρτη μεγαλύτερη γαλακτοκομική εταιρεία ε, στον κόσμο, μεγαλύτερο ε, παραγωγό βιολογικού γάλακτο στον κόσμο. Θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα επίση διασφάλιση ποιότητα, το Arla Garden, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα διατροφική ασφάλεια, περιβάλλοντο και ζωική ευημερία. Έχουμε 75 γαλακτοκομικές εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιε Εκτό Ευρώπη, ε, Θεωρούμε ότι η διατροφική αλυσίδα και όλε οι όλες οι πρέπει να πληρούν σοβαρέ και αυστηρέ προδιαγραφές για να υπάρχει το υψηλότερο επίπεδο διατροφική ασφάλεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η, ο μεγαλύτερη, η αγορά, το 25% ε, ολόκληρου του εισοδήματό μα. Όμω το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μόνο αγορά, είναι και το σπίτι μα. Είναι σπίτι 2.700 Βρετανών γαλακτοκομικών των ε, γαλακτοκόμων ε, και των οικογενειών τους και 3.500 υπαλλήλους ε, Εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, 70% του εισοδήματο των εσόδων του, Ευρωπαϊκού, του, συγγνώμη, της, του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται σε γάλα από του γεωργού μα που κάνουν και την επεξεργασία. Περίπου 160.000 τόνοι γαλακτοκομικών προϊόντων έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 24.000 από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι στην περίπτωση σκληρού Brexit μπορούμε να περιμένουμε 2,7 δις κιλά γάλακτος να μην φτάνουν στο Εμένο Βασίλειο ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να, να βρεθεί λοιπόν μια νέα αγορά, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ε, μια κατάσταση που θα κάνει το εμπάργκο στη Ρωσία να φαίνεται παιχνιδάκι. Σκληρό Brexit θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση στους γεωργούς μας, στην αργοδομιστικότητά μας και στον παγκόσμιο γαλακτοκομικό τομέα. Προσπαθούμε λοιπόν να πληρώσουμε την υψηλότερη δυνατή τιμή για το γάλα μας και να υπάρχουν βιώσιμες θέσεις εργασίας ε, στα αγροκτήματα, ειδικότερα στις περιοχές υπαίθρου, να υπάρχει το πιο ελεύθερο δυνατό εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον Brexit. Ενώ προσπαθούμε να σεβαστούμε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς, που είναι κάτι κρίσιμο για τη βέλτιστη χρήση των, ε, ε του γάλακτος των ιδιοκτητών μας και της διατροφικής αλυσίας. Αν δεν υπάρξει ελεύθερη εμπορική ε, συμφωνία σύντομα, θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε για τη νέα ε, κατάσταση στην αγορά. Με το πιο ελεύθερο δυνατό εμπόριο σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, ε, εννοούμε εμπόριο χωρίς δασμολογικά και μη δασμολογικά ε, εμπόδια. Τώρα, να εστιάζουμε στη διατροφική ασφάλεια, ασφάλεια του τροφίμου σε σχέση με τον Brexit. Με μη δασμολογικά ε, εμπόδια εννοούμε ε, διοικητικό βάρος σε σχέση με το εμπόριο, αλλά ε, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον θα πρέπει να υπόκειται στην νοσιακή νομοθεσία ή τέλο πάντων στο ισοδύναμό της σε θέματα ζωικής ασφάλειας, κτηνιατρικών ε, φαρμάκων ε, ζωικής ε, ευημερίας. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μεταγραφή το, της, ενος, της ενωσιακής νομοθεσίας που ισχύει τώρα στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της, του, νομο, του νόμου αποχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να εξασφαλίζονται τα, οι σωστές προδιαγραφές. Αυτή τη στιγμή ε, η κατάσταση είναι κάπως αβέβαιη. Ε, πάντως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η κυβέρνησή του θέλει να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο θα ισχύει στο μέλλον πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική εμπορική συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου εξασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια των τροφίμων θα είναι ισοδύναμη σε αυτή που ισχύει τώρα η δική μας αξιολόγηση για μετά το Brexit είναι η εξή. Είναι προφανές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρεται ε, για τους καταναλωτές του με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν τα κράτη-μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε σωστές προδιαγραφές ώστε να υπάρχει βέβαια και μια ανταγωνιστικότητα στις τιμές. Οι καταναλωτές ούτε οι λιανοπολιτές και τα οικονομικά δεν, έχει κανένα, δεν έχουν κανένα νόημα ε, στις διεθνείς επιχειρήσεις ε, αν δεν υπάρχει ε, κανένας, καμία εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. Και αυτό τουλάχιστον εμείς στην Arla Foods έτσι το βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν στις τάσεις που υπάρχουν εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ενωμένο Βασίλειο μία τάση κοινή. Θέλουν ασφαλή ε, προϊόντα και ένα πλαίσιο νομοθεσίας και αρχές που να το επιτρέπουν αυτό. Θέλουμε να υπάρχει μία τάση ε, σε σχέση με προσανατολισμένη προς την ενωσιακή προσέγγιση, οπότε θεωρούμε ότι τάσεις αυτές θα διατηρηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν υπάρξουν χαμηλότερε προδιαγραφέ από ό,τι αυτέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Ο συνεταιρισμό μα εστιάζει συνεχώ στη βελτίωση τη ασφάλεια των τροφίμων αλλά και των τροφίμων, μια ε, ισχυρή εσωτερική αγορά ώστε να μπορούν ε, οι γεωργοί να μετακινούνται μεταξύ των συνόρων. Δεν είναι μόνο το η μεγαλύτερη αγορά, είναι και το σπίτι μα και για να βελτιώσουμε τι δεξιότητε του εργατικού δυναμικού μα διασυνοριακά, θέλουμε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη η εμπορική συμφωνία με, την με σεβασμό τη ακαιρεότητα ιστορικής αγοράς. Υπάρχει ένα ισχυρό σημείο αφετηρίας, οι τάσει μεταξύ ε, των δύο πλευρών δείχνουν ότι θα, λογικά θα παραμείνει έτσι. Κατά τη γνώμη μου αποκλίνουσες προδιαγραφέ ασφάλεια των τροφίμων φαίνεται να είναι πάρα πολύ μικρό κατά τη γνώμη μα, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πρέπει οι προδιαγραφέ αυτέ να είναι αναπόσπαστο τμήμα τη μελλοντική μα εμπορική συμφωνία. Όσον αφορά τώρα τον πληθωρισμό, Εντάξει, προφανώ θα υπάρχει μια ισορροπία και πάλι κάποια στιγμή στι αγορέ, αλλά θα υπάρχει α πούμε ε, τα 2,7 δι κιλά γάλακτο που δεν θα πηγαίνουν, ε, δεν θα μεταφέρονται πια από τη μία πλευρά στην άλλη, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα μεσοπρόθεσμα και στι δύο πλευρέ. Το σκληρό Brexit θα δημιουργήσει πρόβλημα στου αγρότε μα, πρόβλημα στου ε, καταναλωτέ λόγω των τιμών και πρόβλημα στι αγορέ και ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχετε στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Σα καλώ λοιπόν Κάτι να υπάρξει μεγαλύτερη και ε, πιο ελεύθερη, η καλύτερη και πιο ελεύθερη εμπορική συμφωνία με μη δασμολογικά ούτε δασμολογικά εμπόδια ώστε να υπάρχει μια νομική ασφάλεια που θα ε, ε, είναι ισοδύναμη με αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή που είμαστε μέλη του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σοντεύης είναι επόμενη από το WITCH, στρατηγική σύμβουλος. Ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω εδώ σε αυτή την ακρόαση. Καταρχάς θέλω να σας εξηγήσω το WITCH, αν δεν ξέρετε τι είναι. Είμαστε μια ανεξάρτητη ένωση καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χρηματοδοτούμεθα από τις πωλήσει πληροφοριών και φυλαδίων που ε, παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές και είμαστε και μη πολιτικοποιημένοι και ανεξάρτητοι. 1,5 εκατομμύρια μέλη και υποστηρικτέ έχουμε. Είμαστε μεγαλύτεροι ενό καταναλωτών στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε ουδέτεροι ε, και μείναμε και ουδέτεροι στο δημοψήφισμα. Ο στόχο μα όμω είναι τώρα η καλύτερη δυνατή έκβαση για του καταναλωτέ από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Στη δέκα τη παρουσίασή μου θα εστιάσω σε τρία ζητήματα κυρίω. Πρώτα απ' όλα, μια επισκόπηση κατάσταση. που βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το πλαίσιο και την ασφάλεια. Έπειτα θα δούμε κάποιες προκλήσεις, κάποιες ευκαιρίες ε, που προσφέρει το Brexit και το τρίτο θα είναι κάποιες προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ξεκινώ λοιπόν ε, σε ό,τι αφορά το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ στενά ήταν συνδεδεμένοι για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζαν ε, την ευρύτερη πολιτική τροφίμων ε, και υπήρξε ένα πλαίσιο το οποίο εξελίχθηκε με βάση διάφορα αισθήματα που μας απασχόλησαν. Είχαμε την όσο των τρελών αγενλάδων, της διοξίνης, ε, το κρέας αλόγου και διάφορα άλλα. Και θεωρούμε ότι το πλαίσιο που υπάρχει είναι κατάλληλο, εξυπηρετεί το σκοπό του. Φυσικά έχουμε τον κανονισμό ε, για τα τρόφιμα που είναι υπό αναθεώρηση στο πλαίσιο του REFIT. Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να τηρούμε. Πρώτα απ' όλα σαφείς ευθύνε αναφέρονται ποιε είναι οι ευθύνε των επιχειρήσεων για την ε, ασφάλεια των τροφίμων. Οι δημόσιες αρχές βέβαια έχουν και αυτές ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για την προστασία των καταναλωτών. Επίση, ε, αναφέρεται το μοντέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αφορά την ανάλυση κινδύνων, που είναι τελείω διαφορετικό σε σχέση με το μοντέλο που εφαρμόζουν άλλε χώρε και είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτό το μοντέλο. Οι βασικέ πτυχέ που ήθελα να τονίσω εδώ είναι η ανεξαρτησία ε, των εκτιμήσεων κινδύνου. Ναι, αναγνωρίζεται η ανάγκη να υπάρχει ανεξάρτητη επιστημονική συμβουλή που θα τεκμηριώνει τη λήψη αποφάσεων, αλλά δεν θα πρέπει το μόνο στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων και βέβαια υπάρχει περιθώριο για ε, άλλους ε, θεμητούς νόμιμους παράγοντες που θα δουν τα θέματα της καλής μεταχείρισης των ζώων και πολλών άλλων στοιχείων που έχουν να κάνουν με τη θέμα των τροφίμων και βέβαια η αρχή προφύλαξη στενά σχετίζεται με όλα αυτά τα θέματα όταν έχουμε να κάνουμε με ανασφάλεια δικαίου. Η δημόσια υγεία είναι το πρώτο. Αν υπάρχουν κίνδυνοι, ρίσκα, ε, δεν τους ξέρουμε όμως πόσο σοβαροί είναι αυτοί κίνδυνη, παρόλα αυτά πρέπει να προστατεύσουν του καταναλωτές. Αυτό είναι ε, το σημαντικότερο. Έχουμε επίσης δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλιση των Τροφίμων, την ΕΦΣΑ πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητοι φορείς. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν, γιατί η ΕΦΣΑ είναι ανεξάρτητη και από τα πολιτικά συμφέροντα και από τα επιχειρηματικά. Και αυτό πρέπει να παραμείνει όταν θα αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν επίση νομοθετήματα για τους ε, μεταλλαγμένου οργανισμούς, για ισχυρισμού υγεία κτλ και τα πρόσθετα τροφίμων και διάφορα. Αλλά έχουμε επίση τον κανονισμό για του επισήμου ελέγχου ε, που προσδιορίζει του ελέγχου που θα πρέπει να γίνονται από τα κράτη-μέλη. Αλλά και η Κομισιόν ε, έχει ένα ρόλο. Πριν υπήρχε εκτινετρική υπηρεσία, τώρα στη ΓΔ ΣΑΝΤΕ υπάρχουν οι φορεί που ελέγχουν ε, την εφαρμογή τη νομοθεσία. Και σε σχέση με τον Brexit θα πρέπει να φροντίζουν οι φορεί αυτοί, οι τρίτε χώρε να συμμορφούνται Προ τι ενωσιακέ απαιτήσει και νομοθεσία. Υπάρχει ένα άλλο, ε, μάλλον υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί συντονισμού που είναι το σύστημα κρισπροειδοποίησης προειδοποίηση, για τρόφιμα, ζωοτροφέ και ένα άλλο σύστημα ε, ανταλλαγή πληροφορών πάρα πολύ σημαντικό ε, τελευταία τέθηκε σε ισχύ και έχουμε και συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για τις εισαγωγές ε, στο Ρότερνταμ ή στα Βρετανικά λιμάνια για να γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια απόρριψη φορτίου και να έχουμε συντονισμένη προσέγγιση. Κοινέ παρόμοιε οι προκλήσει μα λοιπόν και έτσι θα συνεχίσει να, ε, να γίνεται. Είχαμε περιπτώσει στη λιτεριά στον αποτρόφημα, το θέμα του καμπυλοβακτηρίου, ε, χημική ρήπη, ε, πώς θα τους ρυθμίσουμε. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι κοινά προβλήματα και βέβαια και η αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και να από αυτά φυσικά είναι η κλωνοποίηση των ζώων. Ποιες είναι τώρα οι ευκαιρίες. Το λέω έτσι με επιφυλακτικότητα γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η μελλοντική σχέση η Ένωση Ενωμένου Βασιλείου και από αυτή τη σχέση θα εξαρτηθούν και οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι. Από το κατά πόσον δηλαδή θα έχουμε εμπορική συμφωνία και τι θα προβλέπει για τη σχέση μας και σε ποιο βαθμό θα υπάρχει ευελιξία ή όχι για το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να μπορεί να παρεκκλίνει από το σημερινό πλαίσιο της Ένωσης. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι τι θα γίνει με τη μελλοντική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου για τα τρόφιμα και την κτηνοτροφία και τι γίνεται με την κοινωνική πολιτική. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε κοινέ πολιτικές Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών ε, αυτό θέλει να προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, όπω και αν έχει ισχυρού δεσμού μεταξύ υγεία, γεωργία και πολλών άλλων στοιχείων που άπτονται τη πολιτική τροφίμων και τώρα καλύπτονται από διάφορα τμήματα Υπουργείων και άλλου φορεί. Επίση, άλλη ευκαιρία είναι όσο ε, θα αναθεωρούμε τη γεωργική πολιτική, να δούμε αν μπορούμε να ευθυγραμμίσουμε κάποια κίνητρα, δηλαδή παραγωγικότητα, περιβαλλοντική στόχη, ποιότητα τροφίμων, ασφάλεια. Ένα από τα βασικά ζητήματα σε εθνικό επίπεδο είναι πώς θα ενισχύσουμε το καθεστώ επιβολή νομοθεσία που αντιμετωπίζει πρόβλημα, γιατί πιέζονται οι τοπικέ αρχέ αυτή τη στιγμή, ή είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα να αντιμετωπίσει τι προκλήσει που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αν είναι πιο πολύπλοκε εμπορικέ σχέσει, για παράδειγμα. Επίση, θα πρέπει να δούμε τομεί που μπορούμε να ενισχύσουμε τι ρυθμίσει. Και το θέμα είναι πώ θα ε, προσαρμόσουμε κάποια πράγματα, αν μα δοθεί δυνατότητα, όχι όμω ε, άρδιν να αλλάξουμε την κατάσταση. Απλά ό,τι έχει μείνει ατελείωτο, ισχυρισμοί υγεία, προφίλ συστατικό, ε, ηχνηλασιμότητα και κάποια ζητήματα που άπτονται τη επισήμανση και το ετικετοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ουσιαστικά το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει την προσέγγιση για υψηλά πρότυπα ποιότητας ασφάλειας, προστασίας και υγείας. Αυτό δεν πρέπει να διακυβευτεί. Και βέβαια η μελλοντική σχέση, τι φύση θα έχει, αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις διάφορες ε, αποκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν και μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους. Προκλήσεις, τρεις είναι οι βασικές. Ε, το πρώτο είναι ότι η Βρετανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία όλα τα νομοθετήματα. Και αυτό να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμω υπάρχουν κάποιε υπερχειριστικέ πτυχέ που πρέπει να λυθούν το συντομότερο δυνατόν. Τι θα κάνουμε με την αξιολόγηση κινδύνων, τι θα κάνουμε σε σχέση με την ΕΦΣΑ, με κάποια δίκτυα τα οποία βασίζω, στα οποία βασιζόμαστε για τον έλεγχο και την επιβολή της νομοθεσίας προ όφελο και των δύο πλευρών είναι συνεχιστή η συνεργασία. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν το συντομότερο δυνατόν. Σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου, πολλά θέματα αφορούν τι εθνικέ δυνατότητε που θα πρέπει να δημιουργήσουμε, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέου θεσμού ε, αντιγραφή αυτών που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα υπάρξουν αλληλεπικαλύψει και ποια είναι και τα ζητήματα που ε, βλέπουμε στο χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων και συνθήκη. Θα μεταφερθούν σε εθνική νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο για να έχουμε υψηλού επίπεδου προστασίας ε, και των ανθρώπων και των καταναλωτών, αρχή προφύλαξης. Αυτά θα πρέπει να παραμείνουν ως αρχές και στο ε, μελλοντικό δίκαιο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, τη μελλοντική στον Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση έχει πει σε μια λευκή βίβλο για την εμπορική πολιτική ότι θα προωθήσει υψηλά πρότυπα, αλλά πρέπει να φροντίσουμε. Αν ξεκινήσουμε διαπραγματεύσει ε, για συμφωνίε με άλλε χώρε που έχουν τελείω διαφορετικά επίπεδα προστασία και ασφάλεια καταναλωτών, είπα για παράδειγμα, ένα στου έξι Αμερικανού δηλητηριάζεται από τρόφιμα ε, και Ένωση 66 στη Βρετανία κάθε χρόνο με βάση τα πρότυπα των οργανισμών τροφίμων κτλ. Άρα δεν θα πρέπει να χαμηλώσουμε τα δικά μας ε, πρότυπα. Επίσης η δέσμευση των καταναλωτών θα είναι κάτι σημαντικό για το ποιε είναι οι αποδεκτές μέθοδοι παραγωγής στο μέλλον. Οι καταναλωτές έχουν ανησυχίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια αλλά και άλλα ζητήματα. Θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν οι καταναλωτές. Και το τελευταίο που θέλω να πω έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Πέτερ για την πρόσβαση και τι ε, προσιτές τιμές. Δεν πρέπει να υπάρχουν τριβές στο εμπόριο θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά και να δούμε τι σοκ μπορούμε να αποφύγουμε. Δεν θα πρέπει καταναλωτές ή επιχειρήσεις ε, να ε, μειώσουν τα πρότυπά τους, ε, να δοθούν κίνητρα για υποβάθμιση των προτύπων και για απάτες. Προτερότητες λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό είναι το καταληκτικό κομμάτι της παρουσίασής μου. Θα τα δούμε στις διαπραγματεύσεις. Τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να είναι στο επίκεντρο πρέπει να παραμείνουν υψηλά πρότυπα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουμε ε, οι αρχές αυτές να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο. Πρέπει να ενισχύσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την επιβολή της νομοθεσίας και το καθεστώς που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε ευκαιρία να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τα πρότυπα και την ασφάλεια και να περιορίσουμε τις ε, διατροφικές ασθένειες. Επίσης θα πρέπει για την εμπειρία, τεχνογνωσία ε, και τα δίκτυα τα σχετικά να τα ενισχύσουμε. Και σε διεθνές επίπεδο όταν μιλάμε το Επιτροπικό Τεξαλιμεντάριους ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει να Κόντεξ ε, ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει ε, να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Αυτό θα είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Η δε αλυσίδα τροφίμων γίνεται επίσης πιο πολύπλοκη και παγκοσμιοποιημένη και αυτό πρέπει να το λέμε υπόψη. Ευχαριστώ και θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας με τα χαρά Thank Τώρα, Έρωτα Catch the eye. Κύριε Τέιλορ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τους δύο ομιλητές. Ήταν ενδιαφέροντα όσα μας είπαν. Έχω μια ερώτηση για τον ε, κύριο Κάρλσον. Εάν έχουμε hard Brexit και αν επομένω ισχύσουν και εφαρμοστεί δίκαιο γίνουν για τα γαλακτοκομικά εφαρμοστεί του ΠΟΕ, πώς θα επηρεαστούν, τι επιπτώσεις θα υπάρχουν για τους κοινωνικούς παραγωγούς. Ιδίω εκείνοι οι οποίοι κάνουν κάποιο είδου διέλευση και, εξάγουν μέσω του ε, Ηνωμένου Βασιλείου. επίση υπάρχει κάποιο σχέδιο για το ε, τι θα γίνει στην περίπτωση ακριβώς του hard Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να υποβάλουμε τρεις ερωτήσεις και μετά απαντήσεις. Ευχαριστώ τους δύο μιλητές μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, θα μπορούσα να ρωτάω και να συζητήσουμε όλη μέρα, λέει η κυρία Όμως πιέζει ο χρόνος. Έχουμε κάποια προϊόντα τα οποία τα εισάγει το νούμερο βασίλειο, μερικά επιστρέφουν και είδαμε εκείνη την εικόνα με το μωρό που έχουμε αυτό το παιδικό γάλα που μπαίνω βγαίνει στο νούμερο Βασίλειο και εάν ε, έχουμε την παραγωγή στο νούμερο Βασίλειο έχουμε προς την Ένωση εξαγωγές άρα εκεί θα πέσουν οι συναλλαγές θα μειωθούν και εκτός από τα κατατοκομικά έχουμε και άλλα τα οποία θέλουν ακριβόχρονη παράδοση και οπότε άμα κλείσουν τα σύνορα τι θα γίνει όσον αφορά τη μεταφορά με φορτηγά. Έτσι θα γίνει με φορτηγά, έχουμε αρκετά για να περνάνε από τον Τόβερ στο Καλέ. Έχουμε αρκετούς οδηγού φορτηγών. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τον καταναλωτή ε, γιατί υπάρχει σχετική μέρη στο νούμερο Βασίλειο πολύ καιρό. Οπότε για μου, τι εγγύη σα έχουν δοθεί στι συνομιλίε με την κυβέρνηση όσον αφορά την ετικετοθεσία, την προστασία των καταναλωτών, ε, όσον αφορά τα είδη διατροφή, τι υπάρχει κάποιο είδου πλάνο ταχεία ανταπόκριση όταν πια δεν θα ανήκει στην Ευρώπη ε, το νούμερο Βασίλειο και ιδίω αν γίνει κάποιο είδου απότομη ε, έξοδος. πόσο καιρό θα πέρασει ούτως ώστε να συγκροτήσουμε κάποιου είδου ε, ρυθμιστικούς οργανισμούς και αρχές. Um, uh, και εγώ και εγώ να ρωτήσω όπως και οι προλαλήσαντες, λέει ο κύριο Μπράνεν. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει από του μεγαλύτερου θεσμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον μετά το Brexit το περιβάλλον όσον αφορά τα είδη διατροφής θα είναι μεικτό. Μικτό εννοώ ότι θα έχουμε πολλές μεθόδους αντιμετώπισης και οι πλουσιότεροι θα αγοράζουν ε, ε, είδη διατροφής που θα παράγονται στην χώρα γιατί θα είναι καλύτερη η ποιότητα και τα στάνταρ παραγωγής. Όμως ένα σωρό κόσμος ο οποίος έχει χαμηλό εισόδημα δεν έχει άλλη επιλογή. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αγοράζει φτηνά τρόφιμα και αν πρόκειται για ε, Brexit, ε, τότε θα αρχίσουμε να εισάγουμε ε, φτηνά τρόφιμα. Και κάποιοι από τους stories λένε ότι εάν υπάρχει περιβάλλον ελευθέρου εμπορίου θα βγαίνουμε στην παγκοσμία αγορά και θα αγοράσουμε φτηνότερα τα φυτά. Ε, και τότε ο κόσμος θα μπορεί να πληρώνει λιγότερα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι φτηνότερα τρόφιμα ε, πολλές φορές δεν ε, λαμβάνει υπόψη καλό μεταχειριστών ζώων στην παραγωγή, ε, ούτε είναι πάρα πολύ θρεπτικά αυτά τα τρόφιμα και επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουμε ασφάλεια ποιότητα στα στάνταρ παραγωγής για να έχουν προβλήματα ιατρικού χαρακτήρα. Οπότε για πέστε μας την άποψή σας, τι λέτε, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως σενάριο λέμε για φθηνότερο τρόφιμα, αλλά ορισμένοι ε, θα αγοράζουν φθηνά τρόφιμα ε, γιατί δεν θα έχουν άλλη επιλογή. Οπότε θα μεγαλώσει το κομμάτι της αγοράς ε, για τα φθηνά τρόφιμα. Ε, και να, ποιο είναι το μειονέκτημα που θα προκύψει, τι συμφωνούμε, τι όχι. Ε, ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Εσείς. Α, ο κύριος Κάλσεν. Όπως προαναφέραμε, το Ηνωμένο Φασίλειο έχει έλλειμμα στην παραγωγή γάλακτος. Και στην αλυσίδα ε, παραγωγής και στην αλυσίδα προμήθειας. Οπότε και εξαρτώμεθα, εξαρτάται τέλο πάντων από τις εισαγωγές καλακτοκομικών. Αν είναι σημαντική σχέση με την Ιρλανδία για την προμήθεια τσένταρ, το οποίο εισάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και άλλα προϊόντα που εισάγονται από την Ευρώπη. Και το 25% των γεωργών στην Αγγλία μπορούν να παράξουν περισσότερο γάλα αλλά δεν υπάρχει ευρύτερα παραγωγική δυνατότητα και γι' αυτό λέμε ότι από πλευράς καταναλωτή θα πάρει χρόνο μέχρι ότου υπάρξει παντού στο Μένο Βασίλειο ικανή παραγωγή και στη βιομηχανία επεξεργάζονται τα σχετικά σενάρια. Όμως υπάρχει τόση ευαιότητα που είναι δύσκολη η αδίποτε κίνηση. Καμία εταιρεία δεν θα κάνει επενδύσεις στο νούμερο Βασίλειο όταν δεν ξέρουν τι θα απογίνει και τι δασμολογική ή άλλη φραγμή θα υπάρξουν. Τώρα όσον αφορά το γάλα και τα τρόφιμα για μωρά, δεν ξέρω το σύνολο του τοπίου. Δεν ξέρω τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας, αλλά από πλευράς γαλακτοκομικών δεν επαρκεί η παραγωγή μας και θα εισάγονται αυτά τα είδη. Τώρα όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, μια που έχω το λόγο, θεωρώ ότι ενδεχομένως υπάρχει ο κίνδυνος οι καταναλωτές και οι λιανοπολιτές να βελτιώσουν τα στάνταρ. Και έτσι διαφοροποιούμενοι να έχουν και ψηλότερα στάνταρ και φθηνότερες τιμές. Βέβαια υπάρχει ένα σενάριο έλλειψη των γαλακτοκομικών. Οπότε τότε έχουμε εισαγωγέ φθηνών ειδών που να τίθενται σε εμπορία. Ε, γι' αυτό λέμε κι εμείς ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν νομοθετικές εγγύσεις για τα στάνταρ και την ποιότητα και έτσι να προστατευτούν οι καταναλωτές. Ή πρόεδρος για ε, να απαντήσω και εγώ στις δύο πρώτες ερωτήσεις. Όσον αφορά την εξασφάλιση εγγυήσεις από την κυβέρνηση, τι λέει η κυβέρνηση. Δεν προτίθεται να υποβαθμίσει τις εγγυήσεις για την υγεία των καταναλωτών όσον αφορά τα στάνταρ. Όμως, λεπτομέρειες δεν έχουν συζητηθεί, δεν έχουν εξηγηθεί στην πράξη όλα αυτά, πώς θα γίνουν. Και όπως είπα και στην εισήγησή μου, λέει η κυρία Ντέβης, υπάρχει νομοσχέδιο, θα περάσει από τις δύο βουλές και έτσι θα αναπαράγουμε θα αναπαραγάγουμε τέλο πάντων την κοινοτική νομοθεσία. Αλλά πρέπει να γίνει πρώτα αξιολόγηση κινδύνων, υπάρχουν θέματα εφαρμογής νομοθεσίας. Όλα εξαρτώνται από την σχέση με την Ένωση που θα διαμορφωθεί. Έχουμε υπηρεσία για την προτυποποίηση από όλα αυτά τα μελετά. Θα δούμε, θα κάνουμε επιστημονικές επιτροπές, θα συνεργαστούμε με τις κοινωνικές υπηρεσίες όπως η ΕΦΣΑ. Αυτά όλα τα θέματα πρέπει να λυθούν το συντομότερο, να ξεκαθαριστεί. Τι συνεργασία θα υπάρξει. Τώρα όσον αφορά το σενάριο για τα φθηνά τρόφιμα που θα εισαχθούν, ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτό το σενάριο ποτέ δεν θα γίνει πραγματικότητα. Ήδη, λόγω του ότι έχει πέσει η λίρα, έχουν ανέβει τιμέ. Και θα πρέπει να καλύψουν τις ανησυχίες των καταλωτών για την ακρίβεια και να υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια νομοθετικά ελάχιστα για την διατροφική ασφάλεια, για την ποιότητα, να ξέρει ο καταναλωτή ότι αυτό που νομίζει αγοράζει πραγματικά το αγοράζει. Και τέτοια στάνταρ. Αυτές οι αρχές είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν πρέπει να θυσιαστούν στο βωμό της τιμολογιακής πολιτικής. Ναι, λένε ότι έχουμε τα δικά μας ε, στάνταρ για όλους. Ε, αφού έχουμε, ας συνεχίσουν να ισχύουν. Και όσον αφορά τις φτηνές εισαγωγές, ο κόσμος έχει συνηθίσει να έχει την επιλογή. Βέβαια υπάρχουν κάποια εκπτωτικά σούπερ μάρκετ, χαμηλές τιμές, ε, και εκεί πέρα είναι αναμενόμενο να υπάρχουν χαμηλότερα στάνταρ εξαγυρίζουμε. Άρα στο θέμα της εφαρμογής θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο το κράτος να υπάρξουν ουσιαστικοί έλεγχοι και να μην έχουμε ε, λόγω άνων νόδου τιμών ε, και συναφείς απάτες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Έτερος, Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Πίτερ, στη συνέχεια των όσων μας είπες, είναι σαφές το τι θα ισχύσει στο κρατικό μου στην Ευρώπη των 27. Αλλά τι θα κάνουν οι ευρωπαϊκοί φορείς σε σχέση με την ενεργοποίηση του άρθρου 50. Θα έχουμε στρεβλώσεις λόγω του hard Brexit. Θα πρέπει να μην μπλοκαριστεί η χώρα. Υπάρχουν ευθύνε για να εξασφαλιστεί αυτό. Να μην έχουμε αποπληθωρισμό στις τιμές, να μην έχουμε υπερβολική προσφορά σε σχέση με την Ιρλανδία. Για πες μας για τους Ευρωπαίους γαλακτοπαραγωγούς. Λέγονται πολλά όσον αφορά το τι θα απογίνει το σύνορο στην Ισλανδία. η Δημοκρατία της Ολλανδίας ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Θα πρέπει να προσεχωρήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά προς ε, την λύση του ζητήματος και θέλω να ακούσω την απόψη σου. Άλλος, λέει ο Πρόεδρος, έχει κάτι να ερωτήσει. Επιστρέφουμε στους εισηγητές. Έχετε το λόγο. Κάλτσα. Α, ξέχασα να απαντήσω για το τι θα γίνει στο Καλέ. Στον προηγούμενο γύρο απαντήσω. Έχουμε 6.500 containers δικά μας που κυκλοφορούν τα Ιρλανδίας και Αγγλίας. Υπάρχουν ε, εντελεχής τελωνική έλεγε Αυτό θα πρέπει να δούμε και να αποφύγουμε την κυκλοφορική συμφόρηση των φορτηγών στα σύνορα. Ε, αυτό είναι θέμα ουσιαστικό. Και να δούμε και με τις τρεις χώρες τι θα γίνει και να είμαστε αποτελεσματικοί. Τώρα για την ερώτησή σας του σενάριου του hard Brexit. Και τι θα γίνει όσον αφορά τον ΠΟΕ και τα 2.500 ε, εκατομμυρίων, τι είναι, δισεκατομμυρίων κιλών, τέλος πάντων γάλακτος, τι θα γίνει. Ναι, βεβαίως και θα υπάρξουν επιπτώσεις. Το θέμα το έχουμε επισημάνει. Θα πρέπει αυτό να διατεθεί το γάλα είτε στο εξωτερικό είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε έρθει σε επαφή με πολλές υπηρεσίες αρμόδιες για το τι θα γίνει. Βέβαια, χρησιμοποιήσαμε όσο είχαμε στη διάθεσή μας και τελικά απορροφήθηκαν ομαλά οι συνέπειες του εμπάργου με την Ρωσία. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας και προσαρμογής της παραγωγής από πλευράς ε, παραγωγών. Είναι περίπλοκο το θέμα με την Ιρλανδία. Δυστυχώς εξαρτάται από τις εισαγωγές η Αγγλία και για το τσένταρ και για άλλα γαλακτοκομικά. Να βρεθεί λύση. Εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα ποια θα είναι αυτή η λύση δεν έχω την απάντηση προς το παρόν. Άλλο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε ολοκληρώσαμε όσον αφορά το θέμα τη διατροφική ασφάλεια. Μπορεί να καθίσετε να παρακολουθήσετε τη συνέχεια και προχωρούμε στο επόμενο μα θέμα που είναι το περιβάλλον. Η κυρία Σαρλότ Μπέρντ, λάβει το λόγο από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλτ. Mm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παραστώ εδώ σήμερα. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να πω εγώ είμαι τμήμα του ευρύτερου ακαδημαϊκού δικτύου για το Brexit και το περιβάλλον, με ακαδημαϊκούς κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από ολόκληρη την Ευρώπη που ενδιαφέρονται για τον αντίκτυπο του Brexit, για το Ηνωμένο Βασίλειο και για τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές. Αυτή τη στιγμή οι δραστηριότητες μας ε, χρηματοδοτούνται από το Οικονομικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε αν υπάρχουν ερωτήσει ε, που δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα, υπάρχει ένα ευρύτερο δίκτυο στο οποίο μπορώ να απευθυνθώ για να βρω τι απαντήσει. Αυτό που θα ήθελα να κάνω ε, στο πλαίσιο τη παρουσίασή μου είναι να μιλήσω για του λόγου για του οποίου δημιουργήθηκε η Ενωσιακή Περιβαλλοντική ε, Πολιτική, μία περιβαλλοντική, μία που έχει να κάνει με την εμπειρογνωμοσύνη και ένα λόγο οικονομικό. Είναι κινητήρη η μοχλή για την δημιουργία τη πολιτική που εξηγεί για ποιο λόγο είναι επιθυμητό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί αποτελέσει βασικό σημείο εστίασης περιβαλλοντική, να αποτελέσει ε, βασικό σημείο εστίασης για τη δεύτερη φάση διαπραγματιώσεων για το Brexit. Ε, όταν λέμε περιβαλλοντική πολιτική, ε, όπως είχε πει και ο Κλίντον, είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο πρέπει να υπάρχει πολιτική, είναι ότι είναι διασυνοριακή, οι, είναι διασυνοριακές οι συνέπειες. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μία μία αξιοζηλευτή φήμη ως το βρώμικη χώρα της Ευρώπης και αυτό ήταν, αποτέλεσμα, ήταν αποτέλεσμα της κατακαιρματισμένης ε, προσέγγισης που είχε στα περιβαλλοντικά προβλήματα στην αρχή του, της δεκαετίας του 70. χρειάστηκε να δημιουργήσουν καπνοδόχους για να μπορέσει να φύγει ε, η μόλυνση από ένα συγκεκριμένο μέρος και να πάει αλλού. Ε, βλέπουμε επίση ότι υπήρξε για αυτό το λόγο όξινη βροχή στην Νορβηγία ε, και πολλές φορές έχουμε το ίδιο προβλήμα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τον Καναδά και ε, στον Καναδά από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης για τα υγρά απόβλητα φτιάξαμε πολύ μεγάλους αγωγού που μας επιτρέπουν να φτάσουμε για να απορρίψουμε αυτά τα απόβλητα ε, στη Βόρεια και στην Ιρλανδική θάλασσα. Έχουμε λοιπόν τοπικά ε, προβλήματα μόλυνσης, έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτό εξηγεί για ποιο λόγο οι μη κυβερνητικέ οργανώσει του ΕΒ ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τον αντίκτυπο ε, του Brexit ε, και επειδή εμεί ε, ω χώρα δεν έχουμε πολύ μεγάλη παράδοση και καλή παράδοση περιβαλλοντική προστασία, ήδη από το 1970 έχει υπάρξει κάποια πρόοδο λόγω τη προσχώρησή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αποφάσει που λαμβάνονται εδώ και στο Στρασβούργο έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο ΕΒ και είναι πολύ σημαντικό όπω κινούμαστε σε αυτό το νέο πλαίσιο του ισορροπίου του Brexit, να μην υπάρχει ε, ό,τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην έχει αντίκτυπο αρνητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να δεσμεύεται από όλα αυτά τα πρότυπα που εξακολουθούν να το δεσμεύουν όσο είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο λόγο, εμπειρογνωμοσύνη. Όλο και περισσότερο γνωρίζουμε το περίπλοκο των οικοσυστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε όλο και περισσότερο ότι καταλαβαίνουμε πολύ λίγα για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο τη ίδια συμπεριφορά μα είναι σημαντικό να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες και τους σπόρους για να δούμε κατά πόσο οι τάσεις συμπεριφοράς που υπάρχουν σε μία χώρα ε, ή σε μία περιφέρεια εμφανίζονται αλλού. Για παράδειγμα, είναι η μείωση των εντόμων που καταγράφηκε σε φυσικά πάρκα στη Γερμανία. Τώρα οι εμπειρογνώμονες θέλουν, οι επιστήμονες θέλουν να ξέρουν αν αυτό είναι τμήμα μιας ευρύτερης τάσης και ο μόνος τρόπος να το κάνουν αυτό είναι να δουν τι γίνεται και στις άλλες χώρες της Υπήρου. Πρέπει λοιπόν να μοιραζόμαστε δεδομένα μεταξύ μα. Μόνο μέσω τη ανταλλαγή δεδομένων και τη εμπειρογνωμοσύνη μπορούμε να καταλάβουμε τον αντίκτυπο τη ανθρώπινη συμπεριφορά ε, στη φύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μια πλατφόρμα για αυτέ τι ε, ανταλλαγέ απόψεων και μου φαίνεται ότι είναι επιθυμητό το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν γίνεται να έχει και πρόσβαση σε χρηματοδότηση για να μπορεί να συνεχίσει αυτή η, ε, η συνεργασία ο βασικός ε, κινητήριος μοχλός περιβαλλοντικής πολιτικής ένωσης ε, ήταν ε, να μην υπάρχει περιβαλλοντικό dumping ώστε να έχουν όλες τις, τα ίδια πρότυπα όλες οι χώρες. Στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε ήταν η αρχή της συναπόφασης ε, γιατί πολλές από τις περιβαλλοντικές οδηγίες και κανονισμοί είχαν εγκριθεί στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Υπάρχουν πολύ καλοί οικονομικοί λόγοι για να απαιτείται από το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει τα ίδια πρότυπα στο Ηνωμένο, στο, μετά το Brexit για να μπορεί να ε, έχει εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τι ίδιε προδιαγραφέ, α ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια παράλληλη ισοδύναμη νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα παραμείνουν περίπου στο ίδιο επίπεδο. Υπάρχει όμω μια τάση απόκληση μακροπρόθεσμα και αυτό έχει να κάνει νομίζω με το ε, κοινωνικό κεκτημένο. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια πράσινη γραμμή ε, στι διαπραγματεύσει όσο προχωρούν ακόμη και για τους περιβαλλοντικούς νόμους που εγκρίθηκαν υπό τις περιβαλλοντικές διατάξεις της συνθήκης ε, που δεν αφορούν υποχρεωτικά τον ανταγωνισμό ή την ενιαία αγορά, Ξακολουθεί να υπάρχει αντίκτυπος για τον ανταγωνισμό ένα, μια, χώρα, ας πούμε, που κάνει, μια χώρα που κάνει αγρανάπαυση βρίσκεται σε, ε, ε, ε σε οικονομική, οικονομικά μενοκτική θέση σε σχέση με μια άλλη χώρα που δεν το κάνει. Ε, το να, υπάρχει, λοιπόν, να υπάρχουν κοινοί κανόνες διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, και από οικονομικής απόψεως αλλά και από απόψεως οικοσυστημάτων. Τελείωσα λοιπόν τώρα με αυτά τα τρία ε που ανέφερα προηγουμένως. Μερικά ακόμη πράγματα θα ήθελα να πω παρόλα αυτά. Πρώτα απ' όλα το κομμάτι το νομικό. Γενικώ είναι αποδεκτό ότι η νομοθεσία της Ένωσης είναι σαφέστερη και έχει πιο μακροχρόνιες προοπτικές και στόχους σε σχέση με την αντίστοιχη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό που ακούμε συχνά στο Ηνωμένο Βασιλείο είναι ότι η διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία δίνει ένα ευρύτερο ε, πλαίσιο ε, στο οποίο μπορεί να ε, επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά ε, το Brexit, όμως ε, δεν τηρείται τόσο αυστηρά η διεθνής νομοθεσία πάντοτε και συνήθως έχει χαμηλότερα πρότυπα. Κάτι, κάτι λοιπόν το οποίο σημαίνει ότι το επιχείρημα αυτό εγώ το βλέπω με κάποιους συνδυασμούς. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, εδώ υπάρχει ένας τομέας ε, στον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοστάτης, όμως υπάρχουν σοβαρές, ε, σοβαροί κίνδυνοι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τελευταίες ημέρες ε, προχώρησε σύντομα όσον αφορά το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων. Πώς θα μπορέσει τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτύχει τους στόχους τους όσον αφορά τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου αν δεν είναι μέλο μέλος του ETS και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τη δημολόγηση του άνθρακα και των μελλοντικών αγορών. Αυτό είναι κάτι για το οποίο η ε, υπεύθυνη λήψη αποφάσεως ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδιαφέρονται πολύ και ανησυχούν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, πρέπει να ανησυχεί γιατί θα επηρεάσει τη δυνατότητά της να επηρεάσει τους στόχους του στον τομέα αυτό. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με την διπλωματική εμπειρογνωμοσύνη και την πολιτική του Ηνωμένου Βασίλου. Επειδή είχε πρωτοστατήσει για το κλίμα, μπόρεσε να αναπτύξει κάποια εμπειρογνωμοσύνη στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων και διπλωματία, η οποία σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι ε, εκλαμβάνεται πολύ θετικά από του Ευρωπαίου εταίρου. Όπω πηγαίνουμε λοιπόν Προ λοιπόν προς τον Brexit, η συνεργασία είναι σημαντικό να συνεχίσει και αυτή η διπλωματική εμπειρογνωμοσύνη και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεχίσει επίση. Τρίτο σημείο, ισορροπία των πολιτικών στο Συμβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ε, και για την κλιματική πολιτική αλλά και την κοινή γεωργική πολιτική που ε, ε, επιχειρήματα αρκετά φιλικά προς το περιβάλλον. Αν λοιπόν αποσυρθεί το, όταν αποσυρθεί το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χαθεί αυτή η υποστήριξη και συνεπώς να, να φανούν, να, να ακουστούν φωνές πιο σκεπτικές και πιο επιφυλακτικές ως προς την κλιματική αλλαγή ο Πάτρικ εδώ θα μας πει πολύ περισσότερα και με πολύ περισσότερες γνώσεις, αλλά εγώ έχω κάνει συναντήσεις ε, ε, στο πλαίσιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θέμα που επαναλαμβάνεται συνεχώς είναι ότι φοβόμαστε ότι το θέμα του περιβάλλοντος θα ε, ξεχαστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων του Brexit. Εγώ άρχισα την καριέρα μου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως βοηθός πριν κάνω το διδακτορικό μου έχετε πολύ περήφανη ιστορία ε, στη λογοδοσία των ευρωπαϊκών θεσμών και στην ε, προώθηση της περιβαλλοντικής ε, θεματολογίας. Αν τελικά υπάρξει αντίκτυπος, αυτό θα είναι άσχημο και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε ό,τι μπορείτε να μην χαθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του άρθρου 50, να μην πάει πολύ κάτω ως προτεραιότητα η περιβαλλοντική πολιτική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο είναι ο Πάτρικ Engagement, πρόεδρος ε, του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Βόρεια Ιρλανδία. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση προς όλους εμάς. Εγώ σήμερα εκπροσωπώ το Northern Ireland Environment Link, είναι αντιπροσωπευτικός οργανισμός μη κυβερνητικών οργανώσεων από την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά ε, και για τον Ιρλανδικό και περιβαλλοντικό πυλώνα που έχει στην ε, Δημοκρατία της Ιρλανδίας παρόμοια ρόλο και θα εστιάσω στην σημασία του Brexit συνολικά για την Ιρλανδία και θα εκφράσω σοβαρές ανησυχίες για τον δεχόμενο σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον που θα έχει ένα σκληρό Brexit. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά χρόνια καθόριζε το θεματολόγιο των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και χρηματοδοτούσε το περιβαλλοντικό έργο και στις δύο πλευρές των συνόρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ήταν ένα συνεγγυητής των συμφωνιών της Μεγάλης Παρασκευής που υπογραμμίζουν τις πολιτικές ρυθμίσεις που διευθέτησαν το Ιρλανδικό πρόβλημα. Και υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία που και αυτή είναι πολύ σημαντική για την προστασία της κοινή ε, φυσικής κληρονομιάς. Γι' αυτό λοιπόν και καλωσορίζουμε την αναγνώριση στο ψήφισμα του Οκτωβρίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ανάγκη να διασφαλιστούν οι συμφωνημένοι τομείς στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ε, και γι' αυτό χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τη συνεχιζόμενη ε, πολιτική υποστήριξη και το ότι θα τονίσετε πόσο σημασία έχει η συνεργασία να συνεχιστεί για την περιβαλλοντική προστασία και για να αποφύγουμε περιβαλλοντικό dumping. Από ό,τι καταλαβαίνω έχετε ήδη λάβει και ελπίζω να έχετε διαβάσει και το κοινό μας briefing για την περιβαλλοντική ε, συνεργασία που συνοψίζει και προβλέπει κάποιες συστάσεις και έχουμε κάποιες βασικές συστάσεις για το πώς μπορεί να αποφευθεί ένα ε, σκληρό περιβαλλοντικό σύνορο στην Ιρλανδία μετά το Brexit. Πρώτα απ' όλα έχουμε το άρθρο 50, τη διαδικασία αυτή που θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει πλήρω το ζήτημα της διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας δυνάμει της Φωνίας της Μεγάλης Παρασκευής και θα πρέπει το κοινό πλαίσιο τη ενωσιακή νομοθεσία και των πολιτικών και τη μηχανισμοί χρηματοδότηση ένωση να είναι το κεντρικό. Δεύτερον, επειδή η Βόρεια Ιρλανδία και η Δημοκρατία τη Ιρλανδία έχουν κοινά φυσικά ε, περιουσιακά στοιχεία, κοινό αέρα, έδαφος ε, και χλωριτά πανίδα, αλλά και πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα κοινά. Θεωρούμε ότι ε, το νησί της Ιρλανδίας και τα χωρικά του θα πρέπει να θεωρείται μία ενιαία περιοχή, βιογεωγραφική μονάδα. Επίσης, θα πρέπει να διατηρηθεί διασυνοριακή συνεργασία, αλλά να καταπολεμηθεί και ο θέμητος ανταγωνισμός για τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας μετά τον Brexit. Γι' αυτό θα πετηθεί διατήρηση ε, κατά το δυνατό μέγιστης ε, περιβαλλοντικής ευθυγράμμισης της νομοθεσίας, να τηρηθεί και να συνεχίσει να τηρείται το περιβαλλοντικό κεκτημένο. Τέταρτον, πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να εφαρμοστούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί που θα εγγυώνται τουλάχιστον ένα ισοδύναμο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας στη Βόρεια δηλαδή μετά τον Brexit σε αυτό που παρέχει τώρα το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε το σημαντικό ρόλο που παίζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά τη όργανα για την επιβολή τη συμμόρφωση και την εξασφάλιση τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για του πολίτε και την ε, κοινωνία των πολιτών. Αντίστοιχα ισχυροί μηχανισμοί θα πρέπει να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές ε, του συνόρου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε πάλι στο γύρο των ερωταπαντήσεων. Παρακαλώ ποιος θέλει το λόγο να σηκώνει το χέρι του. Madam Um, yes, um... Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Έχω για τον κύριο Κέσμεντ μια ερώτηση. Τι θα μπορούσε να γίνει κάτι γνώμη για να μην φτάσουμε σε μια άβολη κατάσταση ε, όσον αφορά τα σύνορα στην Ιρλανδία. Ίσως θα πρέπει να συγκροτηθούν και θεσμοί, οργανισμοί για να βοηθήσουν, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν λήψεις σε αυτό το επίπεδο στην Βόρεια Ιρλανδία. Κυρία Μαγκίνες, Πρόεδρε, ευχαριστώ και να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι μάλλον δύσκολο, αλλά θα ήταν χρήσιμο να πούμε περισσότερο όσον αφορά αυτό το πρώτο που αναφέρατε, κύριε, δηλαδή τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Είχα πάει στην ΑΦΚΟ και συζητούμε τώρα για το Brexit, για τις δυσκολίες με τα σύνορα στην Ιρλανδία από πλευρά περιβάλλοντο θα πρέπει να αναλυθεί γιατί η Συμφωνία τη Μεγάλης Παρασκευής και η Διασυνοριακή Συνεργασία είναι αλληλένδετα. Και αυτό προβληματίζει όσου ενδιαφέρει το περιβάλλον, γιατί στο θεματολόγιο δεν έχει προτεραιότητα. Ίσως τελικά αποκτήσει προτεραιότητα, αλλά ο κόσμος προβληματίζεται. Μπά και έχουμε για τον Brexit τι εξελίξει που όλοι φοβόμαστε. Τι λύσει δεν μπορούσαν να υπάρξουν. Λάβετε υπόψη τι διαπραγματεύσει. Λάβετε υπόψη το σημείο που βρίσκονται τώρα. Για πέστε μας. Ε, ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε και δίνει το λόγο πρώτο στον κύριο Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τους προσκεκλημένους στο Στασβούργο. Στην επόμενη Ολομελία θα ψηφίσουμε για το Brexit και λέμε ότι δεν έχουμε αρκετή πρόοδο σχετικά αφορά τι διαπραγματεύσεις βάσει του άρθρου 50 και έτσι δεν έχουμε αρχίσει τις διαπραγματεύσεις για το ε, εμπόριο. Βέβαια μπορεί να έχουμε προχωρήσει τι οπότε να έχουμε κάποιε κατευθύνες γραμμέ για τι ε, καθημερινές διαμετεύσει. Αν αυτό το τελευταίο συμβεί, θα πρέπει να δούμε πώ μπορεί να προστατευτεί το πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά κάποια θέματα διασυνοριακά για τη μόλυνση του αέρα, του νερού, για τους οικότοπου, ε, την οδηγία και τα πουλιά. Και ε, θα, πρέπει, για να έχουμε τα ίδια περιβαλλοντικά στάνταρ, να γίνει αυτό το θέμα ε, κάτι που θα προβλέπεται και θα καλύπτεται σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία. Δεν θα πρέπει να φυγεί η Ευρώπη από τυχόν χαμηλότερα στάνταρ της Βρετανίας. Επίσης, τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε συμμόρφωση σε περίπτωση που έχουμε κάποια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, άλλες ερωτήσεις και μετά να ε, έχουμε γύρω Μάλλον πρώτα να απαντήσει και μετά και άλλε ερωτήσει. Κύριο Κέσμεν, ναι, να έχουμε κάποιο είδου ε, καινούριε δομέ, καινούριου οργανισμού. Σχετικά με αυτή την ερώτηση, νομίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ε, νέα δομή στην ε, Βόρεια Ιρλανδία και έτσι να υπάρξει σχετική συμμόρφωση και ε, να καλύψουμε τα, τα κενά, τη αδυναμία που είναι πολύ πιο έντονε από ό,τι στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Να η ευκαιρία επομένω να φτιάξουν τα κακό κείμενα ε, τότε θα πρέπει αυτή η ευκαιρία να μας δώσει, την, να μας δώσει το περιθώριο για να τα καταφέρουμε και να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στο περιβάλλον. Τώρα, όσον αφορά τα διασυνοριακά σώματα, οργανισμούς, τέλος πάντων, δεν μπορώ να σας πω τίποτα δυστυχώς γι' αυτό, αλλά ήδη έχουμε κάποιους οργανισμούς διασυνοριακούς. έχουμε ας πούμε μια, μια οργάνωση που φροντίζει κάποιες, κάποιες λίμνες ε, και από ό,τι ξέρω πάντως το θέμα όντως θα έπρεπε να έχει προσεχθεί περισσότερο. Το πρόβλημα εν μέρη, έγκυται στο ότι τα σύνορα με την Ιρλανδία ακριβώς λόγω αυτών των λιμνών που σας ανέφερα ή τέλος πάντων κάποιων ε, θαλασσίων περιοχών ε, είναι αμφισβητούμενα. Οπότε περιβαλλοντικά οι περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Θα δεν είναι δυνατόν να αδρανίσουμε. Χρειάζεται προστασία. γιατί εκεί έχουμε ένα σωρό επιχειρηματικές δραστηριότητε χωρίς να υπάρχει περιβαλλοντικός έλεγχος. Άρα θα πρέπει να έχουμε καινούργιε δομές στην Βαρελανδία, αλλά ε, να φροντίσουμε οι υπάρχουσες δομές να συνεχιστούν, να λειτουργήσουν οι σχετικές υπηρεσίες και στο μέλλον. Σωστά. Τώρα όσον αφορά τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, μέχρι σήμερα το περιβάλλον δεν έχει καλυφθεί όπως θα έπρεπε από τη Συμφωνία. Ναι, έχουμε συμφωνήσει στα σχετικά με την κοινωνική πολιτική, αλλά τελικά τόσα χρόνια η συνεργασία στα θέματα του περιβάλλοντος ε, απέκτησε σημασία και έχουμε πολλά έργα και προγράμματα που τρέχουν εν μέρη λόγω της ενίσχυσης και της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα για την ειρήνευση από τα ειδικά κοινωτικά προγράμματα από προγράμματα όπως το Live, το Interreg, που έχουν βοηθήσει πολλές ε, πραγματικές προσπάθειες και οπότε όλες αυτές οι ευκαιρίε και αυτή η χρηματοδότηση θα πάψει ή θα συρρυκνωθεί μετά το Brexit. Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα με την περιβαλλοντική συνεργασία και με τη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη Βορειοελλανδία και στην Ιρλανδία. Συμφωνώ με την κυρία Μαγκίνες. Δεν είναι υψηλή προτεραιότητα το περιβάλλον και για αυτό και θέλαμε οπωσδήποτε να έρθουμε σήμερα και να το θέσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε για το πρόβλημα, γιατί είναι σημαντικό. Έχει επιπτώσεις αυτό για όλους μας, για την ατμόσφαιρα, για το νερό. Ε, βέβαια, θα πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα και όσον αφορά πληροφόρηση, όσον αφορά λύσεις, ε, πασχίζουμε να βρεθεί αυτή η λύση. Το πρόβλημα αυτό με τα σύνορα δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι, είναι σχεδόν ε, αδιέξοδο το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε soft σύνορα και ταυτόχρονα αυτό να ε, συμβαδίζει με, την Ευρωπαϊκή, με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, με την Τελωνιακή Ένωση. Αυτά φύγει το Νούμερο Βασίλειο. Πάρα πολύ δύσκολο να παρακάμψουμε το πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάπου θα υπάρχουν βέβαια σύνορα στην Ιρλανδία και θα υπάρξουν βέβαια επιπτώσεις και σίγουρα οι επιπτώσεις για το περιβάλλον θα είναι αρνητικές όταν έχουμε αυτά τα σύνορα τα, hard σύνορα όπως το λέμε. Η κυρία Μπέρντ. Για να απαντήσω τον κύριο Τέιλορ για το τι μοντέλο, τι πρότυπο θα ισχύσει. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι είναι δικητικά αποτελεσματικό και φιλικό στο περιβάλλον και τι είναι πολιτικά εφικτό. Οπότε από πλευράς διοικητικής ε, αποτελεσματικότητας αλλά και για το περιβάλλον θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει να κατοχυρώσει το κοινωτικό κεκτημένο, αλλά αυτό δεν μου φαίνεται πιθανό, γιατί δεν θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα Άλλου είδου συμφωνία θα πρέπει να κλείσει. Αμοιβαία αναγνώριση προτύπων, ισοδυναμία, κάποιο είδου οργανισμό θα πρέπει να συγκροτηθεί και να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει ότι το Ενωργασίλειο συμμορφώνεται με ό,τι συμφωνήθηκε. Και να δούμε αν όπω προχωρούν οι διαπραγματεύσει, αν θα καταλήξουν σε κάτι τέτοιο. Βέβαια, αν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει, γιατί προ παρόν έχουν κολλήσει. Ο κύριο Κέισμεντ. Να προσθέσω το εξή. Ρώτησε ο κύριο Τέιλορ για τι δεσμευτικέ εμπορικέ συμφωνίε. Από ό,τι ξέρουμε, οι κοινοτικές οδηγίες και συγκεκριμένα η οδηγία για τους οικοτόπους και για τα πτηνά, η οδηγία πλαίσιο έχουν επιπτώσεις για το περιβάλλον όπως η οδηγία για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος. Δεν ισχύουν αυτές, αυτά τα νομοθετήματα στην συμφωνία και για τη συμφωνία με την Νορβηγία. και δεν επηρεάζεται το εμπόριο παρόλα αυτά. Επομένως, εμείς θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα ισχύσει με το ημέρο Βασίλειο για οποιαδήποτε δεσμευτική εμπορική συμφωνία που θα γίνει στο μέλλον με την Ένωση. Ευχαριστώ, λέει κύριε Βαλέα. Άλλες ερωτήσεις, κύριε Μπίρντα. Μπίρντερ, μάλλον. Άκουσα τι είπατε για μηχανισμούς ε, εφαρμογής και μας είπατε προηγουμένως για το ότι υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής διεθνώς. Αν επομένω ε, αποχωρήσει η Βρετανία ε, δεν είμαι ουδέτερη, εγώ είμαι κατά του Brexit και αγώνα. Αν αποχωρήσουμε επομένω, τι θα γίνει δύναμη του διεθνούς δικαίου. Θα είμαστε τρίτη χώρα τι θα γίνει με την εφαρμογή. Και κατόπιν των όσων συμφωνηθούν στις διαπραγματεύσεις, βέβαια στις διαπραγματεύσεις δεν είναι προτεραιότητα το περιβάλλον. Και από ό,τι λέμε εδώ στο Κοινοβούλιο, θα πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον να μην παραμεληθεί στην συμφωνία ε, δεν μπορεί να είναι όλα μονόδρομος όσον αφορά την εφαρμογή. Και για τυχόν παραβάσεις θα συρθεί από την Ένωση το Μνήμα Βασίλειο στο Ευρωδικαστήριο. Τι γίνεται επομένω για αυτά τα ζώα, τι γίνεται με το νερό, τι γίνεται με την ατμόσφαιρα, τι γίνεται με, το, με, με την εμπορία ε, των αγρίων ειδών. θα πρέπει να δεσμευθεί το Βασίλειο ότι θα συμμορφωθεί προς το Εθνές Δίκαιο. Μόνο μόνο δούμε. Για πέστε μας τη γνώμη σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπίρτελ. Ο κύριος Τάνς. Και έχουμε ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και σήμερα για τις 4.30 είναι θέμα η Ιρλανδία, οπότε θα φύγω να πάω εκεί. Υπάρχουν πολλά σενάρια για το πού οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις, φόβοι κλπ. Πόσο σημαντικό είναι να δούμε τις επιπτώσεις για το περιβάλλον εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Και ποιο αντίλογο υπάρχει για αυτού που λένε ότι όχι, σενάριο κατάπτωση των διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει. Χαίρομαι που στι 4.30 έχουμε αυτή τη συμφωνία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Γιατί θα πρέπει να συζητείτε περισσότερο και στο σπίτι, στο, συγγνώμη, στην πατρίδα μα. Νομίζω ότι τώρα μην έχει προσεχθεί το περιβάλλον. Είναι ντροπή. Έχετε δίκιο, καθηγητά. Γιατί θα έπρεπε περιβαλλοντικά να ε, λαμβάνει την υπόψη ενιαία η Ιρλανδία, ενιαία ενίσως. Επομένως και οι περιοχές αυτές τις ακτές να θεωρηθούν οικοσύστημα. Βέβαια και όλοι οι το ίδιο. Επομένως έχουμε κάποιο σενάριο που να έχουμε βελτίωση της κατάστασης τελικά Τώρα όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθερών εμπορίου, ε, αυτές απλώνονται μέσα στον χρόνο. Ε, και επίσης παίρνει χρόνο για να συναθούν πώς να περιμένουμε, όπως λέτε με Βασίλειο, ότι θα πάρει 7-8 μήνες η σχετική συμφωνία. Εντάξει, μπορεί να πάρει 7 μήνες, μπορεί να πάρει 7 χρόνια ή 17 χρόνια, αλλά πόσο σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να στείλει ένα μήνυμα ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το περιβάλλον, να προβλέπει στάνταρ για το περιβάλλον ισοδύναμα, τουλάχιστον ισοδύναμα και αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η κοινή γεωργική πολιτική ήταν μια μεικτή ευλογία για το περιβάλλον. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζει καλά η Επιτροπή αυτή. Αν μιλάτε, μιλήσετε σε περιβαλλοντολόγους, θα σας, πει ότι, ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι η κατάλληλη για αυτό που θέλει να επιτύχει. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ε, δεσμεύεται πια ούτως ή άλλως από την κοινή γεωργική πολιτική και μου φαίνεται κάπως δύσκολο να το πω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το αποδέχομαι, αποδέχομαι ότι υπάρχουν ενδεχομένως ε, κάποια ωφέλη εκτός κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες πιστεύετε ότι είναι οι μεγαλύτερες νίκες για το Ηνωμένο ε, Βασίλειο και ε, για τα ε, νησιά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Κυρία Burns, σας ευχαριστώ πολύ όσον αφορά το μηχανισ... τους μηχανισμούς επιβολής. Εξαιρετική ερώτηση ε, για την οποία και εγώ και άλλοι λαμπροί δικηγόροι δεν έχουμε απάντηση για το, το θέμα της επιβολής, του μηχανισμού ε, επιβολής για τις τρίτες χώρες, επειδή είμαστε σε μια μοναδική κατάσταση αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο τι σημαίνει δεν υπάρχει κάτι έτοιμο που να μπορούμε να πούμε, α, ωραία, θα πάρουμε αυτό το μηχανισμό και θα τον χρησιμοποιήσουμε αμέσω, ειδικότερα όταν το Ηνωμένο Βασίλειο λέει ότι δεν θέλει να υπόκειται στη δικαιοδοσία ε, της ε, ε, ε, του δικαστηρίου της ΕΦΤΑ ή ε, του δικαστηρίου της Ένωσης σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ένας άλλος μηχανισμός όσον αφορά τα μεταναστευτικά είδη και την, το λαθρεμπόριο άγριων ειδών. Ε, προφανώς υπάρχουν και κάποιες διεθνείς ε, συμφωνίες ε, που δεν αποτελούν δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι συμφωνίες παρέχουν αρκετά καλά πρότυπα ώστε να μπορούν να επιτρέψουν στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου να προχωρήσει επιτυχώς. Όσον αφορά τα σενάρια βελτίωσης περιβαλλοντικών προτύπων, νομίζω ότι αυτό ήταν η μία ερώτηση. Εννοείται εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι. Βεβαίω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, για τον οποίο η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σήμαινε ότι θα καταστούν χειρότερα, χειρότερα τα πρότυπα. Υπάρχουν ευκαιρίες διαθέσιμες να πιέσουμε για πιο φιλόδοξα πρότυπα και το βλέπουμε αυτό ε, στη Σκοτία και στην Ουαλία για παράδειγμα. Οι πολιτικές είναι πιο φιλόδοξες σε σχέση με την κλιματική αλλαγή από ε, αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου σε εθνικό επίπεδο. Σε μία μελέτη όμως που εγώ και κάποιοι συνάδελφοι από το, το, Πανεπιστήμιο ε, του Queens και του East Anglia προσπαθήσαμε να δούμε, να συμπεριλάβουμε αυτούς τους παράγοντες. Δηλαδή τι θα γίνει αν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα διέπεται πια από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίσαμε να δούμε πώς μπορεί να σχεδιαστεί η νομοθεσία η οποία παραδοσιακά ήταν λιγότερο ευρωπαϊκή σε άλλους τομείς εκτός από την περιβαλλοντική πολιτική και καταλήξαμε, και μου έκανε εντύπωση αυτό, στο ότι οι περιβαλλοντικές πολιτικές ήταν πολύ χαμηλότερες και ε, ήταν πολύ χαμηλότερης ε, προτεραιότητας, ενώ οι οικονομικές πολιτικές πάντοτε κέρδισαν. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού ε, ε, Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με τα άγρια είδη, για παράδειγμα, ε, πολλοί κόσμος θα σας πει ότι καλύτερα να ισχύουν οι ενωσιακοί νόμοι γιατί είναι σαφέστεροι και πιο εύκολο να εφαρμοστούν ενώ οι ντόπιοι νόμοι είναι πολύ πιο δύσκολοι, πολύ πιο δυσνόητοι και επίσης ε, πάντοτε οι οικονομικές ε, ε, πολιτικές τις καπελώνουν. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν γιατί να μην υπάρξουν πιο φιλόδοξες πολιτικές περιβαλλοντικές. Ιστορικά, ανεξαρτήτως της κυβέρνησης, δεν είναι κάτι το οποίο έχει κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν μπορέσαμε πάντοτε να πιέσουμε περισσότερο με πιο φιλόδοξα περιβαλλοντικά ε, ε, ζητήματα, ενώ το κάναμε με την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Κάτι ακόμη. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πιο σταθερές, πιο σταθερά πλαίσια πολιτικών και πιο μακροπρόθεσμο ε, χρονικό ορίζοντα. Ε, οπότε υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια κυκλοθυμικότητα σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου λόγω τη αλλαγή των κυβερνήσεων για παράδειγμα όταν δεν θα δεσμεύεται πια από την, από την ενωσιακή πολιτική. Εν πάση περιπτώσει πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ε, ως νίκη αν καταφέρουμε να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε μια πολιτική περιβαλλοντική ε, πιο φιλόδοξη ε, και πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε τοπικές συνθήκες. Υπήρξε μάλιστα και μία έκθεση για τον αντίκτυπο για τα αγροπεριβαλλοντικά πρότυπα και εξετάσαμε συγκεκριμένα αυτά τα ζητήματα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, Κάποιο από το RSPB είπε ότι όταν πρόκειται για το Brexit ε, οι απειλέ είναι γνωστές και πραγματικές ε, και οι ευκαιρίε είναι απλώς θεωρητικές. Και το λέω αυτό δυστυχώς και σε σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική γιατί υπάρχουν πολύ γνήσιες ανησυχίες σε σχέση με τη χρηματοδότηση ε, υπό την, τον τρέχοντα διακανονισμό Σκοτία, Ουαλία παίρνουν πολύ χρηματοδότηση από την κοινή γεωργική πολιτική. Δεν είναι βέβαιο όμω ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη χρηματοδότηση αυτή μετά τον Brexit. Επίση, τι αρχέ ε, θα υπάρξουν σε σχέση με τη γεωργική πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, η Επιτροπή Περιβαλλοντικού Ελέγχου ε, είπε ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι θα, υπάρξουν, θα, υπάρξουν κάποια, θα υπάρξει κάποια δημόσια χρηματοδότηση. Όμως αν ρωτήσετε τους αγρότες, εκείνοι προτιμούν την έμφαση στην ασφάλεια τροφίμων. Το θέμα λοιπόν είναι ε, πώς θα οργανωθεί, πώς θα σχεδιαστεί η νέα κοινή ε, ε, γεωργική πολιτική. Για να τονίσω αυτό που είπε η Σαρλότ, συμφωνώ απολύτως για αυτό που είπε για τη μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική. Ενδεχομένω είναι μια τεράστια ευκαιρία να βελτιώσουμε τα περιβαλλοντικά πρότυπα, συνειδητοποιώντα παράλληλα ότι υπάρχει αυτή η ευκαιρία. Υπάρχουν όμω και φόβοι, σοβαροί φόβοι, πραγματικοί φόβοι, ότι αν πιέσουμε τους ε, ε, ιδιοκτήτες γης και τους ε, γεωργούς πάρα πολύ, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους και εμείς εξαρτώμαστε πλήρως από αυτούς ώστε να υπάρχει ένα περιβαλλοντικό όφελος στην Ήπεθρο. Δεν μπορεί να γίνει με διαφορετικό τρόπο, πρέπει να γίνει μέσω αυτών των ανθρώπων που έχουν τη γη στην κυριότητά τους και υπό τη διαχείρισή τους. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τη γεωργία αλλά και παράλληλα να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζουν οι γεωργικές δραστηριότητες χωρίς αυτό να είναι επιβλαβές για το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν ε, να, ε, να εξευρεθεί μια ισορροπία και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τα για τα υπόλοιπα ερωτήματα τώρα, ως προς τη συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής, ναι, δεν την, ε, δεν την χάνει ιδιαίτερη ε, προσοχής, είναι σαφές αυτό. Όταν ήρθα εγώ στις Βρυξέλλες για να μιλήσω σε ανθρώπους που συμμετέχουν στις, διαπρα... στις διαπραγματεύσεις, όλοι γνωρίζουν την συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και τον αντίκτυπό του. Όταν πάει κανείς στο Λονδίνο να μιλήσει στον κόσμο εκεί, είναι σαφές ότι έχουν έτσι μια πολύ ε, δικόνα του περί τίνος πρόκειται. Και να σας πω την αλήθεια αυτό είναι πολύ θλιβερό. Ελπίζω ότι θέτοντα το θέμα εδώ ε, και σε άλλα φόρα, ελπίζουμε μπορεί να θέσουμε το θέμα τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής γιατί νομίζω ότι είναι ενδεχομένω κάτι που μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη συμφωνία ε, μια ε, αποχώρησης του Ηνωμένου Βασίλειου Καλής Κοιτάξτε, ε, εμείς έχουμε τεράστιο... Υπάρχει πολύ κοινό έδαφος ως προς τα μεταναστευτικά πτηνά. Έχουμε γύρω-γύρω θάλασσες όπου υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία σχεδόν ε, των πάντων ε, και μιλώ κυρίως για ε, τα είδη των νυχθείων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κοινά στοιχεία, υπάρχουν όμως και τεράστιες διαφορές ε, στη Χλωρίδα και στην Πανίδα μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας ε, ε, και φυσικά διαφορετικά από την υπηρετική Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν διαφορές, αλλά νομίζω ότι η διαχείριση βάσει κοινών προτύπων και κοινών ρυθμιστικών μηχανισμών είναι ένα θετικό βήμα και βασικό θέμα αν θέλουμε να προχωρήσουμε γιατί διαφορετικά τα είδη μπορεί να, υποχρεώνουν, ε, να υποφέρουν στη μία, ε, στην επικράτεια όπου υπάρχει ε, λιγότερο καλή νομοθεσία. Και θα ήθελα επίσης να πω ε, ότι αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να στείλει ένα μήνυμα για τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τη διατήρηση των προτύπων αυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά από το Brexit, ε, εγώ πραγματικά θα το θεωρούσα αυτό πάρα πολύ ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σημειώσετε, ως πρόεδρος, τα σχόλια του κ. Κέισμεντ για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με το θέμα που συζητούμε σήμερα. Δηλαδή να ενημερωθούν οι διαπραγματευτές για τον Brexit και ιδίως ο κύριος Παρνί. για τις ε, ε, για τα όσα είπε, επειδή εγώ εκπροσωπώ τη Βορειολανδία, τη μεθοριακή περίοδο. Πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ νοχλητικά, πάρα πολύ απογοητευτικά. Γιατί δημιουργείται μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια για τις σχέσεις ε, και στο εσωτερικό του νησιού και μεταξύ των νησιών των δύο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως παρατήρηση. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για το τι ευκαιρίες έχει το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Όμως, τι προτίθεται να κάνει με το εμπόριο το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω λάβει μεικτά μηνύματα για το αν θα διατηρηθούν ε, ή όχι τα πρότυπα, οι κανονισμοί, αν θα είναι αυστηρότεροι, ψηλότεροι, χαμηλότεροι κτλ. Δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλάμε για τη γεωργική πολιτική και αν δούμε χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία που δεν υπάρχουν υποστηρικτικά συστήματα, υπάρχουν και εκεί πολύ σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Άρα δεν έχει κάποια πολιτική για τη γεωργία ε, βρει ε, το τέλειο, ε, την τέλεια λύση για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα. Και έχουμε και την πολλαπλή συμμόρφωση και τις πληρωμές. Αν ακούν τη συζήτηση οι αγρότες, θα τους καλούσα να προσέξουν αυτό που είπε ο κύριος Κέσμα, ότι χρειάζεται υποστήριξη για τη διατήρηση αυτών των δημόσιων αγαθών οι αγρότες και εκτινοτρόφοι πρέπει να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Θα ακούσουμε και από τον Επίτροπο Χόγκαν αύριο τι πιστεύει για ε, τις ανάγκες μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και τι θα πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της πολιτικής. Πρόεδρος. Φυσικά και τα αποτελέσματα της ακρόασής μας θα, θα τα διαβιβάσουμε στους διαπραγματευτές. Αυτό το είπα και στην αρχή, αλλά δεν ήσασταν μάλλον εδώ. Ένα ερώτημα από την κυρία Γκέρλινγκ τώρα. Ευχαριστώ. Όχι ένα, δύο-τρία ερωτήματα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει πίεση από στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς που είμαστε μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ούτε καν θέλουμε να το πιστέψουμε κάτι τέτοιο. Γιατί δεν θεωρούμε να υποβαθμιστούν τα πρότυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υπάρξει αντίστοιχη πίεση στην Ένωση. Αλλά υπάρχει αυτό το εδεχόμενο ε, και για παράδειγμα αν το Ηνωμένο Βασίλειο αποσυρθεί από τη συμμόρφωση στο ΡΙΤΣ, αυτό θα έχει επίπτωση εδώ, στις 27, γιατί μιλάμε για την αγωνιστικότητα. Πολύ σωστά, είπατε Σάρλοτ, ότι η ανταγωνιστικότητα ήταν η βάση του, ε, της πρώτης δέσμης νομοθετημάτων για την νέα αγορά. Πολύ ισχυρό εργαλείο. Και για το φράκινγκ, την υδρορογμάτωση, που θα βλέπουν τι κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο τα άλλα κράτη-μέλη. Και δεν νομίζω να γίνει αλλού βέβαια. Θα μπορούσε όμως να γίνει, αν ξαφνικά είχε πρόσβαση σε πολύ φθηνή ενέργεια του Ηνωμένου Βασίλειου. Αυτό θέλω τώρα να το συσχετήσω με αυτά που γίνονται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του άρθρου 50. Το όλο ζήτημα της πρόσβασης στις αγορές. Η συζήτηση δεν έχει επεκταθεί στο τι σημαίνει αυτό και για το περιβάλλον. Ούτε εδώ, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι ποτόθωρο κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας γιατί νομίζω ότι είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα το ότι θα πρέπει μέσα στο πρόβλημα της ε, πρόσβασης αγορές να συμπεριλάβουμε τις περιβαλλοντικές πτυχές. Επίσης, επόμενο ερώτημα. Ένα είδος θεματοφύλακα της περιβαλλοντικής ακαιρεότητας είναι η Επιτροπή μας. Τι θα πρέπει, πιστεύετε, εμείς να πετήσουμε από αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη όλα αυτά τα ζητήματα. Πανεξέταση περιβαλλοντική νομοθεσία και αναθεώρηση ενδεχόμενη. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο. Έχουμε το effort sharing. Γενικώ το αναφέρω, όχι στο πλαίσιο το νομοθετικό σήμερα. Περισσότερε περιβαλλοντικέ ε, ρυθμίσει ε, επιμένουν τα βάρη μεταξύ των 28. Αν βγάλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο τι υποχρεώσει του, τι θα κάνουμε, θα το διαιρέσουμε και θα πάρει ο καθένα ένα κομμάτι κατά πάσα πιθανότητα θα ξανανοίξει όλη η συζήτηση για όλα αυτά τα νομοθετήματα περιβαλλοντικά. Ποια είναι η δική σας άποψη ως προς τις ε, και βραχυπρόθεσμες και πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Τέλος, είναι ένας καθαρός εισφορέας ε, στη χρηματοδότηση των προπολογισμών το ΕΕ. Μιλήσαμε για τους ε, αγρότες και πραγματικά Πολλά λέγονται ότι αυτό θα είναι μια ευκαιρία για το περιβάλλον και για την κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει όμως να μας ξεφεύγει ότι θα μειωθεί πολύ ο προπολογισμό. Μιλάμε για 2-2,5 δις. 3,5 όμως είναι το πόσο σήμερα στο Μήνο Βασίλειο. Δηλαδή η μείωση θα είναι τεράστια. Και αυτό θα επηρεάσει τις ε, χώρες, τις υπόλοιπες, τις 27 χώρες της Ένωσης. Θα με ενδιαφέρει η άποψη και γι' αυτό. Και κάτι άλλο που θα με ενδιαφέρει είναι μην υπάρχοντα στο Μέρο Βασίλειο ω καθαρό ε, χορηγό, ε, χρηματοδότη, ε, ο προπολογισμό Ένωση, τι θα απογίνει, έχουμε την ΕΦΣΑ που στηρίζεται από το γενικό προπολογισμό. Δεν υπάρχουν τέλη που να την υποστηρίζουν. Δεν θα επηρεαστεί. 27 καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να αυξήσουν την αναλογία χωρίς τη συμβολή του Βασιλείου για την ε, οργάνωση αυτή που είναι στην πρώτη γράμμη της πελωτής προστασίας. questions? Άλλες ερωτήσεις. Αφού δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, εσείς πάλι. Θέλετε να αρχίσετε. Um, just, just to start, oh, to start on the για να ξεκινήσουμε από το εμπορικό το οποίο είναι αλληλένδετο με την απορρίθμιση λέει ναι αυτό φοβόμαστε περισσότερο να έχουμε απότομο ή hard Brexit και να μην γίνει κάποια συμφωνία όπως ε, είπαμε και προηγουμένως τότε το Ηνωμένο Βασίλειο οπωσδήποτε θα πρέπει να πάει να βρει άλλους εμπορικούς εταίρους με χώρες που θα έχουν χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Τα είπαμε σε σχέση με τα τρόφιμα. Ε, το ίδιο ισχύει και με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Άρα, Θα να, ότι θα χαμηλώσει ο πύχης όσον αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα, γιατί με χώρες τέτοιες θα έχουμε συμπήξει συμφωνίες. πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει υπάρξει πρόβλημα στην Ιρλανδία γιατί είχε χαμηλότερα πρότυπα η Βορειός Ιρλανδία οπότε ε, μπορούσαν να έχουν πλέον έκτημα είχαν χαμηλότερες τιμές παραγωγής τροφίμων από τη Δημοκρατία της η οποία τώρα θα μπει στον πειρασμό να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν θέλετε να επιβιώσουμε εμπορικά θα πρέπει και εμείς να κατεβάσουμε τον ε, πύχη ακριβώς όπως κάνει και η Βόρεια Ιρλανδία. Ε, τότε θα υπάρξει πίεση και για τους 27. Νομίζω, αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση, ένα σενάριο, αλλά υπάρχει ανησυχία ότι αυτό μπορεί να είναι μια ακουσία συνέπεια. Εάν επιταχυνθούν οι διαδικασίες και τελικά ξαφνικά σχετικά αποχωρήσει το Το βασίλειο. Η Γύρω και μίλησε για το φράκινγκ. Νομίζω ότι υπάρχουν σχέσεις αντίρρησης τη Βόρειο Ιρλανδίας και στην Δημοκρατία τη Ιρλανδία. Μια που υπήρξε από πλευράς ε, κεντρικής κυβέρνησης ισχυρό ενδιαφέρον. Άρα κατά κάποιο τρόπο ε, με τους συμπατριώτες μας έχουμε έτσι ρίξει περισσότερο από ότι με τους γείτονες εμείς στο Μέρο Βασίλειο. Ε, να δώσω τη σκητάλη στην ε, κυρία Μπέρνς. για την πίεση προς ε, απορρίθμιση. Εγώ θα τα πω άλλη οπτική γωνία. Έχουμε ένα κράτος μέλος το οποίο περισσότερο από όλους τους άλλους έχει πιέσει για να υπάρχει απορρίθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έκανε λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο το Δεν θα είναι πια εδώ και αυτό που να πει ότι η πίεση για απορρίθμιση θα χαλαρώσει, θα εξαφανιστεί. Όπως είπε και ο Πάτρικ, θα υπάρξουν συνέπειες για την ε, Ιρλανδία και έμεσα επομένως ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που αναδύεται. Τώρα όσον αφορά πούμε, και για το Ρίτς, θα με εξέπλησε ε, το να αποσυρθεί από το Ρίτς η Βρετανία γιατί κάποια κράτη θέλουν να προσβέσουν στην ευρωπαϊκή αγορά και συμμορφώνονται με το ΡΙΤΣ και ε, το εφαρμόζουν, συμμετέχουν χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε τώρα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Είναι τεράστια αγορά Ευρωπαϊκή Ένωση. 27 κράτη το σύνολο είναι ισχυρότερο από το κάθε κράτος χωριστά οικονομικά. Ε, αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνούν οι διαπραγματευτέ. Και θα πρέπει το περιβάλλον και τα πρότυπα να μην τα ξεχάσουν οι διαπραγματευτές για οποιαδήποτε συμφωνία. Να τα σκεφτούν καλά. Να απαιτηθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσει ισοδύναμη νομοθεσία. Είπατε επίσης και για επανεξέταση της ε, νομοθεσίας σε με το κλίμα. Ναι, θα ξαναμοιραστεί η τράπουλα, αλλά να δούμε τι θα γίνει. Ξαρτάται και από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Σε αυτή τη φάση. Για τον προπολογισμό. Πολύ σωστά το ρωτήσατε. 12% λαμβάνει υπηρεσία περιβάλλοντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια είναι καθορισμόρια στο Ερμηνό Βασίλειο και αυτό θα αντιμετωπιστεί στις διαπραγματεύσει. Πάντα, πάντα ήταν θέμα, τώρα θα είναι πιο σοβαρό. Ότι με το Brexit θα υπάρξει οικονομική, δημοσιονομική ασφυξία. Και θα έχουμε ένα σωρό απρόβλεπτες επιπτώσεις το περιβάλλον θα υποβιβαστεί ακόμη περισσότερο, θα χάσει θέσεις στην κατάταξη των θεμάτων. Έχουμε τώρα δύο συνεργεία το No Deal, κάτι το οποίο το λέγαμε και που ήμασταν προετοιμασμένοι και επίσης υπάρχει και μια εξέλιξη του να έχουμε no deal, απότομο, ξαφνικό και έχουμε άλλα θέματα, χημικές ουσίες, από, απόβλητα, πολλά πολλά που θα είναι καταστροφικά, αλλά θα υπάρξουν και στην την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να προσθέσω κάτι για την χρηματοδότηση της Γεωργίας. Σήμερα η Βόρεια Ιρλανδία λαμβάνει 9% του προπολογισμού για την γεωργία από την Ένωση τριπλάσια πόσο θα έπαιρνε εάν η κατανομή γινόταν με τη βάση του πληθυσμού και τώρα υπάρχουν φόβοι ότι μόνο θα χάσουμε αυτή την ενίσχυση αλλά θα υπάρξουν ακόμα λιγότερα για περιβάλλον και γεωργία από την Αγγλία. Οπότε έτσι η Βόρεια Ιρλανδία θα έχει πρόβλημα επειδή θα βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανησυχίες πολλές γι' αυτό. Σημαντικό. Και έτσι θα έχουν μεγάλο μειονέκτημα οι Γεωργοί στη Βόρεια Ιρλανδία σε σχέση με τους γεωργούς της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. να ξαναγυρίσουμε τώρα στα εμπορικά. Ε, βέβαια, οι μελλοντικέ συμφωνίες θα μπορούσαν άνετα να είναι χτύπημα για την γεωργία μας. Ξέρω δεν είναι το θέμα της συζήτησης, αλλά περιβάλλον και γεωργία είναι θέματα ελέγχοντα. Εμεί είμαστε καθαρός εξαγωγίας γεωργικών προϊόντων. Βόρειος Ιρλανδία προς Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, προτεραιότητες μας διαφορετικές, αλλά σε κάθε συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε φθηνά είδη και θα πρέπει να ε, προσεχθεί αυτό το κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι εξαγωγέ. Ξέχασα κανένα που θέλει να ρωτήσει. Ο κύριος Ντάντς. Σύντομη ερώτηση. Για την καθηγήτρια Μπέρνς. Έχει γίνει κάποια μελέτη για την επίπτωση των IN, επί των INDC σε σχέση με την ε, Συμφωνία των Παρισίων ε, άπαξ και αποχωρήσει το Μένο Βασίλειο ξέρω ότι στη Συμφωνία των Παρισίων ε, ε, εκπροσωπείται χωριστά το Ένω και η Ένωση, αλλά κάτι διάβασα για αυτό που λέτε, δεν θυμάμαι πού. Οπότε θα ψάξω. Και βράχει πρόθεσμα για τα NDC δεν θα υπάρχει συμφωνία. εθνικά καθορισμένη πρόθεση συνεισφοράς. Είναι το INDC. οπότε σαφώς το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί ότι θα πρέπει να δεσμεύεται σε κάποιες εσωτερικές πολιτικές ή αποφάσεις και προσπαθεί ε, να πετύχει τους ε, στόχους για το διοξίδιο του άνθρακος. Να δούμε. Πρόεδρος, καλώς και σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε για τις ερωταπαντήσεις και σας συναδέλφους, και προχωρούμε. Στο τρίτο τμήμα της συζήτησης. Υγεία. Παρακαλώ. Να λάβουν θέση ο κύριος Πολ Λάφιν. Σα ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα για τι ενδεχομένε απειλέ που αναδύνονται όσον αφορά το επάγγελμα, το λειτουργήμα των ιατρών, αλλά και τις απειλές για τους ε, ασθενείς και ε, εγώ ε, δουλεύω στον ιατρικό σύλλογο, BMA είναι τα αρχικά και θα αναφερθώ έτσι στον ιατρικό σύλλογο και ασχολούμαι με τις δημόσιες υποθέσεις, είμαι διαχειριστή δημοσίων υποθέσεων. Τώρα πρώτα απ' όλα μία μικρή εισαγωγή για τον Ιατρικό Σύλλογο, είναι επαγγελματική, ε, επαγγελματικό φορέας και ε, εκπροσωπούμε 150.000 ε, φοιτητέ και γιατρούς καθηγητικότητας σε όλη τη χώρα. 8.000 είναι οι γιατροί οι οποίοι παίρνουν την ειδικότητά τους. Επίσης και προέρχονται από χώρες του ΕΟΧ, ε, Αγγλία, Ουαλία που ψήφισαν υπέρ του Brexit, Σκοτία και Βόρειος Ιρλανδία που ψήφισαν κατά. Είναι μέλη μας. Από τότε που έγινε το δημοψήφισμα, ο Τουρκός Σύλλογος αναλύει ε, την νομοθεσία. Τι προβλέπεται για ε, τις ιατρικές αγωγές στην Ευρώπη. Έχουμε συνεργαστεί με τους εθνικούς ε, ιατρικούς συλλόγους, ούτω ώστε να επικοινωνήσουμε για όλα αυτά. Ευχαριστούμε ότι δώσατε σήμερα την ευκαιρία. Έχουμε επικοινωνήσει και με τις εθνικές κυβερνήσεις, όσες εξπροσωπούνται στη χώρα μας. Πιο σημαντικό τώρα το οποίο έχουν να δημιουργήσουν οι γιατροί και στην Ευρώπη και στην Αγγλία είναι η εργασία αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων. 21.000 είναι οι γιατροί που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 9% είναι το συνόλου των εργαζομένων. Βλέπετε εδώ τα σχετικά νούμερα. Και αυτό το 9,1% αν δείτε τις ειδικότητες το, έχουμε και τον τέταρτον των φαρμακοποιών που στη χώρα μας ήρθαν και προέρχονται από άλλη χώρα. Και το ένα ε, πέμπτο των, ε, των ιατρών και χειρουργών. Να, σε αυτή την φωτογραφία βλέπετε όλο το τοπίο Ιούνιος, 24 Ιουνίου του 16 σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου. Όπως μπορείτε να δείτε, έξι από τους επτά γιατρούς σε αυτή την υπηρεσία πήραν το πτυχίο τους σε άλλη χώρα. Χωρίς την βοήθειά τους και χωρίς το σύστημα υγείας, μάλλον το σύστημα υγείας θα είχε καταρρεύσει. Και δεν έχει ωφεληθεί βέβαια μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο από την αμοιβή αναγνώριση και την ελεύθερη διακίνηση εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες γιατρών εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μία εβδομάδα το μήνα στην Ουγγαρία, στην Πορτογαλία και δύο ε, εβδομάδες στην Ισπανία και έτσι εξασφαλίζεται το ότι η αμοιβαία αναγνώριση θα ωφελήσει όλους, όλα τα συστήματα υγείας. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε έναν Πολωνό ε, γιατρό, ο οποίος εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να εξυπηρετεί στη γλώσσα τους, τους Πολωνούς ασθενείς. Και όταν γυρίσει στη χώρα του θα έχει μάθει όλα τα καλά που έχει το επάγγελμα στην ε, στην Αγγλία. Να, τώρα βλέπετε στη Ρουμανία. Έχει 30 χρόνια εμπειρία κάποιο και έχει χρησιμοποιήσει την εμπειρία του αυτό ο χειρούργος. και επίση έχουμε έναν Ιταλό ο οποίος τώρα εκπαιδεύεται για ειδικότητα στην Γερμανία αλλά εργάζεται στον Ηνωμένο Βασίλειο. Όπου και να αποφασίσει να δουλέψει θα ωφεληθούν οι ασθενείς του από όλες τις δεξιότητες της εκπαίδευσης και σε Γερμανία και σε Αγγλία. Άρα όλοι βγαίνουν κερδισμένοι τώρα. Εάν υπάρξουν περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση, περιορισμοί για το πού μπορούν να δουλέψουν, ε, τότε θα έχουμε ένα πλήγμα για το σύστημα υγείας. Αλλά το, τα στήματα υγείας παντού και στην Αγγλία και στην Ευρώπη. Και κάναμε μια έρευνα τον περασμένο μήνα και ρωτήσαμε τι σημαίνει το Brexit για σας, τι προτίθεστε να κάνετε. 50% δυστυχώς είπαν ότι σοβαρά μελετάμε το να αναχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά να φύγουν από όλη την Ευρώπη και να πάνε Αυστραλία, Ασία, Αμερική και πρόκειται για κάποιους ε, πολύ εξειδικευμένους, αγγλομαθείς γιατρούς. Αυτή είναι η αγορά, ε, για αυτού είναι ένα προστατευμένο περιβάλλον. Να, ένα Πολωνό θα κερδίσει στην Πολωνία 45.000 δολάρια το χρόνο. Ο ίδιος γιατρός Πολωνός στο Ηνωμένο Βασίλειο 140.000 δολάρια και αν αποφασίσει να πάει στην Αυστραλία μπορεί να φτάσει τα 240.000 δολάρια. Να, να, ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία ότι άμα σφίξουν το πράγμα του Ηνωμένο Βασίλειου αυτοί θα γυρίσουν τη χώρα προέλευση. Επίσης, το Brexit είναι σοβαρή απειλή και για την ασφάλεια των ασθενών δεν θα σταματήσει η μετανάστευση και χάρη στην, στο, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένας μηχανισμός ε, προειδοποίησης για όποτε υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Και βλέπετε ότι από τότε ξεκίνησε αυτός ο μηχανισμός, το 2016 Έχουμε την αρμόδια αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει προειδοποιήσει για αυτούς τους συναγερμούς ας πούμε δύο φορές περισσότερο από ότι οι ευρωπαϊκοί αντίστοιχοι οργανισμοί. Και αν αυτός ο μηχανισμός δεν υπήρχε τότε ένας γιατρός που είχε διαγραφεί από το Σύλλογο στην Βρετανία να γίνει χώρα καταγωγή, α πούμε τη Δανία και αυτό θα ήταν απειλή για του ασθενεί διότι θα ήταν διαγραμμένος. Επίσης, πολλή κουβέντα γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για το αυτοί που ψήφισαν για το Brexit κατάλαβαν ότι θα φύγουν από την ενιαία αγορά. Για να πάμε να το προχωρήσουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι κάποιοι, περίπου το 1% κατάλαβε ότι η αποχώρηση από την Ένωση σημαίνει αποχώρηση και από την Ευρατόμ. Ένωση και ενέργεια και αυτό γιατί είναι σημαντικό, διότι η Ευρατόμ διευκόλυνε το να υπάρχει εξασφάλιση ραδιοϊσοτόπων από την Ευρώπη, να χρησιμοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και έχει σημασία για διαγνώσεις και για τον καρκίνο. Άμα επομένω δεν συμφωνηθεί το να μείνουμε εκεί, τι σημαίνει για το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο όταν φύγουμε το Μάρτιο του 19 σε λίγες μέρες θα πρέπει να βρει ραδιοϊσότοπα από αλλού. Γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για μας. Διότι θα έχουμε καθυστερήσεις σε διαγνώσεις, θα έχουμε ακυρώσεις επεμβάσεων και μακροπρόθεσμα και στην Ευρώπη και στην Αγγλία θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία η οποία θα περιοριστεί. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ιρλανδικό πρόβλημα. Προηλία να το έδωσε στην και όσον αφορά την Ιρλανδία είναι 7%, 1,8% στη Βορειοελλανδία και 4,8 στην Δημοκρατία Ελλάδα. Σύνολο περίπου 7. Οπότε θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ούτως να εξασφαλίσουν τις εξηγημένε ιατρικέ υπηρεσίε. Για παράδειγμα, ε, στο Δουβλίνο την ε, πρωτεύουσα έχουμε το μόνο Ινστιτούτο Καρδιολογίας της χώρας για παιδιά και έρχονται εκεί οι ανήλικοι για αγωγή ε, Χωρί να φύγουν στο εξωτερικό. Ε, καταλαβαίνετε πόσο ωφέλεια υπάρχει. Το ίδιο ισχύει και για το London Dairy και εκεί υπάρχει Εκεί επίσης υπάρχει ένα μοναδικό νοσοκομείο που έχει ειδικότητες που δεν υπάρχουν αλλού και, στο Ντόνεγκαλ επίσης εκεί έχουμε καρδιολογικές υπηρεσίες εκεί, για την ε, κομιτεία του Ντόνεγκαλ Αυτά από το Μάιο του 16. 27 ήταν ε, αυτή τον οποίο η ζωή σώθηκε μια που μπόρεσαν να πάνε εκεί. Ε, βλέπετε, είναι θέμα ζωής και θανάτου. Τόσο ομά τίθεται εν κατακλείδη εδώ βρίσκομαι από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου της Βρετανίας δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος των Ευρωπαίων ιατρών. Παρ' όλα αυτά συνεργαζόμαστε στενά με ευρωπαϊκές ε, οργανώσεις ιατρών που εκπροσωπούν γιατρούς και από τις 27 χώρες μέλη. Συμφωνούν μαζί μας και βλέπετε αυτή τη διαφάνεια που είναι, ήταν σε ένα, αυτό πήγε στον κύριο Μπαρνιέ, πήγε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ότι δεν θα πρέπει το Brexit να αποτελέσει απειλή για την υγεία στην Ευρώπη. Παρακαλούμε και εσείς κάντε ό,τι μπορείτε για να μην συμβεί αυτό που φοβόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Virginia Άκα τώρα, που είναι εκτελεστική διευθύντρια ε, MSD και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακοβιομηχανιών και ε, συλλόγων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Νομίζω ότι είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω και να συνεισφέρω στη σημερινή ακρόαση. Και άλλωστε είμαι και η τελευταία μετά από πάρα πολύ παρόμοια μηνύματα που προσπαθήσαμε όλοι να περάσουμε για το μέλλον του Brexit και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, ολοκληρώνουμε τη δουλειά που έχουμε αρχίσει εδώ και χρόνια. Το βασικό μου μήνυμα σήμερα ε, είναι ότι παρά το γεγονός ότι βλέπουμε βασικές προκλήσεις και για τη δημόσια υγεία και για τους ασθενείς, ε, ε, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο λόγω του Brexit. Ε, ε, έχουμε εδώ τους συναδέλφους, είμαστε και εκ μέρους του ΕΦΠΙΑ, εκπροσωπούμε και το ΕΦΠΙΑ. Είμαστε πάρα πολύ αφιερωμένοι στο σκοπό της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη αναστάτωση. Πρέπει όμως να υποστηρίξουμε, να μας υποστηρίξετε και εσείς να προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. Δύο πράγματα θέλουμε να ζητήσουμε. Πρώτον, σε σχέση με την, Ευρωπαϊ... με την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Συνεργασία, θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσει η συνεργασία και ρυθμιστικά πρότυπα ε, και πρακτικές ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων μεταξύ άλλων και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, τα... την παροχή ε, φαρμάκων από την παραγωγή μέχρι την παροχή του στους ασθενείς και επίσης μια μετάβαση ομαλή για να μπορέσουμε να το, πετύχουμε να το αυτό με λογικό τρόπο γιατί μέχρι τώρα ε, από τώρα μάλλον, από τον Νοέμβριο του 2017, ο χρόνος ε, δεν είναι με το μέρος μας. Πρέπει λοιπόν να είναι μια προτεραιότητα που θα γίνει πολύ σαφή στη διαπραγματευτική ομάδα, όπως είπαν κι άλλοι σήμερα στην ε, ακρόαση. Πρέπει να περάσουμε και σε αυτές τις συζητήσεις το συντομότερο δυνατόν, γιατί μέχρι τώρα από την ενεργοποίηση του άρθρου 50 ε, τα τρία τέταρτα της χρονιάς περιμένουμε να γίνει αυτή η συζήτηση και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο για να ε, καλυφθούν αυτά τα ζητήματα. Να σας εξηγήσω λίγο πιο συγκεκριμένα τι θέλω να σας πω. Καταρχάς, να σας ε, κάνω μια απεικόνηση για τον κύκλο ζωής ενός φαρμάκου. Δύο η ώρα, για παράδειγμα, τα 30-40 τελευταία χρόνια επενδύσεων στην Ευρώπη ε, μέσω της φαρμακευτικής νομοθεσίας που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συνεισφορά της Επιτροπής σας έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Φαρμάκων ε, για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη διαδικασία σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη δημιουργία μέχρι την παροχή στον ασθενή ενός φαρμάκου. Ε, εμείς έχουμε συμμετάσχει πάρα πολύ στις επενδύσεις αυτές. Το μερίδιό μας είναι αρκετά σημαντικό σημαντικό, ε, για παράδειγμα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για κλινικές δοκιμές. Επίσης έχουμε και τις κλινικές δοκιμές ε, ε, που έχουν τον Ηνωμένο Βασίλειο Σπόνσορα, 1.500-400 κεντρικά εγκεκριμένα προϊόντα που έχουν, ε, ε, το οποίο, των οποίων κάτοχος άδεια είναι το Ενωμένο ε, Βασίλειο. Θέλουμε να συνεχίσει η συνεργασία και τα αποκεντρωμένα προϊόντα βέβαια είναι χιλιάδες που δεν τα έχω συμπεριλάβει στον υπολογισμό μου. 1.300 προϊόντα τα οποία δοκιμάζονται και ε, παρέχονται, φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο και πηγαίνουν σε ασθενείς ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προς χρήση τους και επίσης τα δεδομένα αυτά προέρχονται από μια έρευνα που έκανε το EFIP ε, ε, φέτος. 45% των μελών της EFIP θεωρούν ότι θα καθυστερούν αυτά τα φάρμακα αν πρέπει να πέσουμε πάλι στους κανόνες του ΠΟΕ και τέλος για τους ασθενείς, και τέλος για τους ασθενείς, σκεφτείτε τον όγκο με τον οποίο έχουμε να κάνουμε για τα διάφορα πακέτα ε, και τις δόσεις ε, που παρέχουμε στα διάφορα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. 45 εκατομμύρια τα οποία τα παρέχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη των 27 ε, βλέπουμε λοιπόν πάρα πολύ σαφώς ε, ότι ήταν σωστή η ολοκλήρωση, αποτελεσματική. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη να την αναιρέσουμε όμως και γι' αυτό ε, πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο την αλυσίδα παροχής, την αλυσίδα διανομής, ε, ε, γιατί ε, μπορείτε να δείτε για παράδειγμα από απόψεων προϊόντων ε, είναι αμφίδρομη αυτή η ροή προϊόντων και αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ παραγωγικό στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, την παραγωγή των σωστών ε, προϊόντων για χάρη των ασθενών. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το εξασφαλίσουμε μέσω του κεντρικού συστήματο ότι όντως θα φτάσουν τα φάρμακά μα στου ε, ασθενείς που, ε, που τα χρειάζονται. Να σας εξηγήσω ας πούμε να, μια απεικόνηση που μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε. Ε, βλέπετε για παράδειγμα ένα ε, φάρμακο για το AIDS. Ε, Βλέπετε λοιπόν τι τεράστιο αντίκτυπο μπορεί να έχει ε, ο οργανισμός ε, ε, φαρμάκων ευρωπαϊκός. Καταρχάς υπάρχει μία ενιαία έγκριση, υπάρχει μία, μία, ένας ενιαίος έλεγχος διανομής και ένας ενιαίος έλεγχος, μια ενιαία παρακολούθηση της ασφάλειας για ένα ενεργό λοιπόν φαρμακευτικό προϊόν όταν πρέπει να έρθει από την Ιαπωνία πρέπει να περάσει από το τελωνίο και πρέπει να περάσει και από, μια, από ένα ρυθμιστικό έλεγχο καταλληλότητος πρέπει να ελεγχθεί και να εγκριθεί για να διατεθεί για χρήση και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν φτάσει λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί εκεί ξεκινά, δεν σταματάει όμως εκεί ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά ε, γίνεται ανάληψη σε διάφορες εγκαταστάσεις, πηγαίνει στην Ισπανία για ανάπτυξη, ε, μπορεί να επανέλθει στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν έχει ολοκληρωθεί για διανομή. Σε αυτή τη φάση ε, διανέμεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της. Σε αυτή την περίπτωση το ενιαίο σύνορο είναι μεταξύ της Ευρώπης και μίας τρίτης χώρας. Αφού θα γίνει το Brexit, ε, προφανώς θα υπάρχουν και καινούργια σύνορα τα οποία θα υπάρξουν στην αλυσίδα διανομής και όπως καταλαβαίνετε ο αντίκτυπος ε, των καθυστερήσεων ε, της παροχής των φαρμάκων θα είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην ΕΦΠΙΑ. υπάρχουν και άλλοι πολλοί σύλλογοι που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί η Medicines for Europe για παράδειγμα η ASGP για την μεταφορά και τη διανομή φαρμάκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρησιμοποιήσαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία για να γράψουμε κατευθείαν στον Μισελ Μπαρνιέ για να μπορέσουμε να τονίσουμε αυτά τα σημαντικά στοιχεία τα οποία σας αναφέρω σήμερα ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει συνεργασία και η ρυθμιστική συνεργασία όλος ιδιαίτερος για να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η σημαντική ανταλλαγή επιστήμης, προϊόντων, υπηρεσιών ε, μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τώρα ε, περιμένουν από εμά να τους παρέχουμε αυτά τα φάρμακα. Κάθε συμφωνία πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει αντίστροφο αποτέλεσμα όσον αφορά την πρόσβαση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, ε, ζητούμε ε, χρόνο για να δούμε τα δικαιώματα των χρηστών για να μπορέσει να συνεχιστεί τουλάχιστον ε, για πάρα πολύ κρίσιμες περιπτώσεις, για έναν ασθενή στην Πολωνία, ένα ένας ασθενής στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην καταλάβει τη διαφορά του Brexit στην κατάστασή του. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Μπορώ να ολοκληρώσω γιατί η διαφάνεια ούτως ή άλλως ε, ουσιαστικά αποκρισταλώνει αυτό που είπα προηγουμένω, ότι η συνεργασία είναι ειπα προηγουμένω, οτι πολύ μεγάλη σημασία και μελλοντικό, οποιοδήποτε μελλοντικό τομέα ε, με μοντέλο συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενωμένου Βασιλείου είναι κρίσιμη σημασία για την παροχή φαρμακευτικών προϊόντων. Θα θέλαμε να σα ζητήσουμε να μα βοηθήσετε ε, καθιστώντα αυτό μια προτεραιότητα για να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, το συντομότερο δυνατόν, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε το στόχο αλλά και με την αλλαγή τουλάχιστον μία περίοδος εφαρμογή μετά από το 2019 χρειάζεται ώστε αυτές οι αλλαγέ στην αλυσίδα διανομής να γίνουν ομαλά, να ξέρουμε ότι θα υπάρχει όντω παροχή των φαρμάκων, είναι δύσκολες περίπλοκες διαδικασίες και περίπλοκα, ε, πολύπλοκε προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Από την άλλη όμως... Ε, ε, αυτό έχει επιτύχει 40 ε, χρόνια συνεργασίας, ε, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον ε, για τα φάρμακα και την διανομή τους. Σας ζητούμε λοιπόν την υποστήριξή σας για να το πετύχουμε αυτό για την ώρα με την αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων. Πραγματικά αφήνουμε τους ασθενείς να αναρωτιούνται και να σκέφτονται μα τι θα γίνει και θα είναι κάποτε έτοιμα τα φάρμακα. Θέλουμε λοιπόν να σας ζητήσουμε την υποστήριξη σε αυτό το σχέδιο που είναι το καλύτερο σχέδιο για το μέλλον των φαρμάκων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος έχει ερωτήσεις, ήδη έχω δύο εγγεγραμμένους στον κατάλογο, ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, δύο ομιλητές. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι με την Φρανσουάσα Γκροστέτ το συζητήσαμε λίγο μεταξύ μας και καλό θα ήταν όλες αυτές οι επιπτώσεις να είχαν ληφθεί υπόψη πριν το δημοψήφισμα για το Brexit διότι έπρεπε να είναι γνωστό ότι θα υπάρξουν προβλήματα στον τομέα της υγείας, προβλήματα για τους ασθενείς. Και τώρα ε, το θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα κάνουμε ώστε να τον λιγότερα αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά συνηγορούν υπέρ ενός ε, ε μια συμφωνίας, μια συνθήκης και όχι ενός σκληρού ε, Brexit. Η κυρία Άκα ε, είπε ότι έχετε ενημερώσει τον κύριο David Davis έχει γίνει γνωστό αυτό το πρόβλημα και για τον Πολ Λάφιν έχω το ίδιο ερώτημα. Έχετε επαφές με τη Βετανική κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά τους ε, υπεύθυνους της διαπραγμάτευσης ε, των, ε, από την πλευρά του Βασιλείου έχουν γίνει κατανοητά αυτά ή θα πρέπει να ακουστεί πολύ πιο ηχηρή φωνή των ασθενών. Και θέλω να σας μιλήσω για την οδηγία σε ό,τι αφορά τη δεσυνοριακή ατροποφαρμακευτική περίθαλψη πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς. Μετά το Brexit τι θα γίνει στον τομέα αυτό. Έχετε κάποιες σκέψεις. Thank you. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ε, πράγματι, ακούγοντάς σας, σκέφτεται κανείς ότι είναι λυπηρό. Ο λαός ε, ήταν αυτός που θέλησε τον Brexit και ο λαός θα υποστεί τις συνέπειες. Βλέπουμε πολύ καλά εδώ ποιε είναι οι ευθύνε των πολιτικών. Αυτό έτσι ήρθε εν παρόδο, αλλά έπρεπε να το πω. Μιλήσατε πράγματι για τους ασθενείς, είναι προφανές και μας εδώ στην Επιτροπή μας ανησυχεί πάντα το θέμα αυτό και τους ασθενείς έχουμε στο μυαλό μας πάνω απ' όλα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τι γίνεται με τις ε, φαρμακοβιομηχανίες, πώς ετοιμάζονται, πώς προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του Brexit. Το Brexit πώς επηρεάζει τις ε, στρατηγικές επενδύσεων ε, των φαρμακοβιομηχανιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μιλήσατε για τι αλυσίδε εφοδιασμού και καταλαβαίνω ότι είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Μέχρι στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο εφάρμοζε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τη διάθεση των φαρμάκων στο εμπόριο για να βρεθεί μια λύση. Μηπω μία συμφωνία μια συμφωνία βία αναγνωριση θα ήταν μια λύση για τα φαρμακά έχουμε συνάψει ως Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες συμφωνίες με άλλες χώρες. Μήπως αυτή θα ήταν μια λύση, τουλάχιστον μια προσωρινή λύση, για να μην έχουμε διακοπή του εφοδιασμού και με όλες τις επιπτώσεις που αυτό συνεπάγεται για τους ασθενείς. Πρακτικά τα ερωτήματά μου, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ακούσουμε την άποψή σας επ' αυτού. Και συμφωνώ με την ερώτηση του Πετελίζε για την οδηγία σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μπορεί να αφορά την Ορβηγία την Ελβετία. Αυτέ οι χώρε ε, εφαρμόζουν αυτή την οδηγία για τη διασυνοριακή ατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μια συνέχεια και με το νούμερο Βασίλειο βέβαια για να γίνει αυτό πάρα πολύ σημαντικέ είναι οι που θα πρέπει να καταβάλει η Βρετανική κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση η Ευρώπη ε, δεν νομίζω ότι θα το κάνει στη θέση του. Πρώτα, σταματήσω με αυτέ πρώτα τι δύο ερωτήσει και θα περάσουμε στην επόμενη. Στον επόμενο γύρο μετά. Να απαντήσετε. Ποιο θέλει πρώτο στο λόγο. Κυριάκα, ευχαριστώ πολύ για την ε, δυνατότητα που μου δίνετε να σας δώσω κάποιε περαιτέρω διευκρινήσει. Ήταν εξαιρετικά τα ερωτήματα και πολύ εύστοχα. Αν είχαμε κάποια επαφή με τη Βρετανική κυβέρνηση η, ο Υπουργό Θεϊκών ε, στον τοπικό τύπο και στο National Times δημοσίευσε μια επιστολή που έλεγε ότι θέλουν να, έχουν συνεργασία με την Ευρώπη για τις ρυθμίσεις και νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθούμε να πιέζουμε την κυβέρνηση και σας εγγυώμαι κύριε Λίζε ότι κάθε ευκαιρία που έχουμε την αξιοποιούμε για να εξηγήσουμε όσο δυνατόν σαφέστερα τις ανάγκες μας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που χρειάστηκε να διευκρινίσουμε με το Υπουργείο του κ. Ντέιβις είναι να καταλάβει ότι για μας, για τον κλάδο το δικό μας και για άλλους που ακούσαμε νωρίτερα στην ακρόαση το θέμα δεν είναι μόνο οι εμπορικές διευθετήσεις, δηλαδή ε, το, οι δασμοί, αλλά τα μήνα δασμολογικά εμπόδια. Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να έχουμε ευθυγράμμιση και συνεννόηση. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Γκροστέτη, την αναγνώριση Είναι οι σχετικέ συμφωνίε σε ισχύ για την Ελβετία, για παράδειγμα, και για τα MRI και τις ε, άλλες ε, έρευνες με τις ΣΥΠΑ, για παράδειγμα. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες για να έχουμε αντίστοιχη προσέγγιση στο θέμα αυτό και νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας εδώ. Και είναι μια ευκαιρία αυτή. Γιατί οι Βρετανικοί φορεί ε, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται αυτή τη στιγμή ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Δικτύου. Άρα από την ίδια αφετηρία ξεκινάμε. Δεν είναι λοιπόν ανέφικτη μια συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν. Και εδώ θα θέλαμε όσο το δυνατόν περισσότερο να υπάρξει σύγκληση. Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι αν ετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε και άλλα σενάρια. Πράγματι, χωρίς ε, αμφιβολία στον δικό μου τομέα και η δική μου εταιρεία αλλά και άλλες εταιρείε ε, ετοιμάζουν ε, προγράμματα έκτακτη ανάγκης. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι έχουν υποχρεώσει. Έχουμε άδειε, έχουμε εγκρίσει εδώ στην Ευρώπη και πρέπει να παράσουμε τα προϊόντα μας. Όμως αναγνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες να γίνει αυτό τόσο σύντομα. Εξού και ζητούμε χρόνο εφαρμογή για να μπορέσουμε να φέρουμε σωστά ε, σε πέρα καθήκοντά μα. Ε, Κύριο Λάφιντ, από το Δόκτωρα Λίζε, αν μιλάμε στην Βρετανική κυβέρνηση, φυσικά και μιλάμε. Εγώ θα συναντηθώ με έναν από του υπουργού ε, του Brexit την Πέμπτη και το μήνυμα ε, είναι πάρα πολύ σαφές από το BMA, την Βρετανικό Ετρικό Σύλλογο. Και όπως καταλαβαίνετε μιλάμε και στην Task Force της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ερχόμαστε σε επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους και λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό αφορά το εργατικό δυναμικό που τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο απόκλησης μεταξύ Βρετανικής κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τους, ιατρικούς, τους ιατρικής. Εάν κάποιο είναι φοιτητής ιατρικής ε, Γερμανό στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2021 μετά το Brexit ε, ε παίρνει πτυχίο, δεν είναι βέβαιο ότι θα αναγνωρίζονται αυτά τα προσόντα ε, αυτοί σπουδών ε, στη χώρα σου μετά το Brexit. Και είναι λάθο, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά η αμοιβή αναγνώριση των προσόντων των επαγγελματικών και των τίτλων σπουδών θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Εμείς το λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ζωές των φοιτητών, αλλά ο μελλοντικό επίσης ιατρικός προγραμματισμός και τα συστήματα υγείας δεν θα πρέπει να τα θυσιάσουμε όλα αυτά. Το δεύτερο που έχει να κάνει με την οδηγία της τη συνορική υγειονομική περίθαλψη, πολύ σημαντικό, τεράστιο θέμα, χαίρομαι Βάσει από ε, ε, του ε, βουλευτέ που εκπροσωπεί το Γιβραλτάρ είναι εδώ στην αίθουσα, γιατί αυτό θα εφαρμοστεί στο υπερπάντη αυτό διαμέρισμα ε, το Βρετανικό που είναι το Γιβραλτάρ. Οι 200.000 ε, εκπατριστέντε μετά το Brexit, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στο Γιβραλτάρ που είναι εκεί 32.000 και να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να συμβεί, δεν είναι βιώσιμο. Γι' αυτό και δεν είναι ο μόνος λόγος, αλλά είναι ένας από τους λόγους που ζητούμε οι Βρετανοί υπήκοπος ε, και εμείς να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως είχαν μέχρι τώρα. Και τούμπαλιν. Ε, και για το δόκτωρα Λίζε ένα άλλο ερώτημα που έθεσε είναι τι γίνεται με τη διασυνοριακή ε, αντιμετώπιση σπάνων ασθενειών. Πράγματι υπάρχουν κάποια δίκτυα που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι πάντα σχετικό όμως με το εργατικό δυναμικό. Αν δεν έχουμε ειδικού, αν δεν έχουμε τις ειδικότητε για αυτά τα δίκτυα αναφορών, αν δεν είναι στελεχωμένα με ειδικού, αυτά τα δίκτυα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και εδώ είναι το θέμα της αμοιβές αναγνώρισης σημαντικό για να παραμείνουν Ευρωπαίοι γιατροί και στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κυρία Πίρντερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες και αυτές οι ομιλίες. Δεν το είπαμε αυτό κάτι διάρκεια του δημοψηφίσματος. Ναι, το είπαμε. Και μας είπαν ε, ότι κάθε φορά που λέγαμε δηλαδή ότι αυτό ε, θα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, μας είπαν ότι φοβόμαστε η κυβέρνησή μας πρέπει να το καταλάβει αυτό. Ελπίζω να το καταλαβαίνει. Πάντως δεν φαίνεται να έχουν την ε, ικανότητα... Τη γνώση ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους και αυτό που ακούσαμε σε σχέση με τα πρότυπα για τα τρόφιμα και για τα ε, φάρμακα. Αυτή η κοινή γεωργική πολιτική, η κοινή ελευτική πολιτική, τα χημικά, τα τρόφιμα, τα πάντα. Όλοι έρχονται σε εμά, ε, Βρετανοί ε, ευρωβουλευτέ είμαστε και έρχονται και μα λένε το καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ο αντίκτυπο, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο βεβαίω πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να ασκήσουμε πιέση στην κυβέρνηση μας στο Ηνωμένο Βασίλειο για να βγει κάτι από αυτό και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι τόσο πολύ που έχουμε αυτή την ακρόαση σήμερα και η υπόλοιπη Ένωση πρέπει να το καταλάβει αυτό. Ακούσαμε ότι γίνονται έρευνες μεταξύ των ε, ιατρών και αν δεν μείνουν στην Ευρώπη υπάρχει περίπτωση να πάνε κάπου αλλού. Είναι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία την οποία πληρώσαμε όλοι προκειμένου να εκπαιδευτούν αυτοί οι άνθρωποι και όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο υπολογίζουμε σε αυτούς. Το θέμα τώρα των μεταγγίσεων αίματος ή των ε, μεταμοσχεύσεων ε, αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Το ερώτημά μου είναι η, ε, επιδοτήσεις για έρευνα, επειδή εμείς είμαστε αποδέκτες τεράστιων ποσών, επειδή έχουμε πολύ καλά ερευνητικά νοσοκομεία. Ήταν πάρα πολύ μάλιστα σημαντική και η δράση που ανέλαβε ε, ο σχετικός ε, σύλλογος για όλα αυτά. Τι θα γίνει, θα αλλάξει αυτό. Αυτή όλη η ειδική ε, οι ειδικευμένοι άνθρωποι πού θα απορροφηθούν, πού θα μετακινηθούν. Επίσης το, η μετακίνηση του οργανισμού φαρμάκων, τον χάνουμε εμείς, τον κερδίζουν οι κάτω χώρες. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Αν τώρα πρώτα εμείς να κάνουμε τις δικές μας αξιολογήσεις φαρμακευτικών προϊόντων, τις ιατρικές αξιολογήσεις, πού θα βρούμε τους ανθρώπους που θα το κάνουν αυτό, ερωτώ. Επίσης, ε, τι, ποια πιστεύει ο μιλητής ε, η ε, πιθανότητα για να, για, να, για να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα να τεθεί ένα αμφιβόλο όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχει περίπτωση εμείς να πάμε να ζητήσουμε φθηνότερες εισαγωγές ε, ε, ε, φαρμάκων από Κίνα ή Ιαπωνία, τέλος πάντων όπου αλλού παρασκευάζονται με χαμηλότερες τιμές και αυτό είναι καλό για την υγεία των Βρετανών. Τι αντίκτυπο θα έχει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ερώτηση για τον κύριο Λάφιν. Άκουσα με ενδιαφέρον τα προβλήματα σε σχέση με την Ευρατών και τις συνέπειες από την αποχώρηση. Τι επιπτώσεις θα υπάρχουν με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί θα πρέπει να απευθυνθούμε σε τρίτες χώρες για τα ενεργά ισότοπα. Επίσης, για πέστε μας, τις επιπτώσεις ε, επί των 27 όταν δεν θα συμμετέχει στην Ευρωτόμ ως μέλος η Αγγλία. Επίσης έγινε κάποια διαβούλευση με το PMA σε σχέση με την ε, Εθνική Αρχή των Μεσανίγειας ε, είναι διαβούλευση για την ενδεχόμενη αποχώρηση των Ευρωτών. Ναι, σε ευχαριστούμε. Ήταν πάρα πολύ ολοκληρωμένες αυτές οι εισηγήσει για τα ζητήματα τα σχετικά με τη, το ιατρικό επάγγελμα του ασθενείς, την νοσηλεία. Και καταλαβαίνουμε πόσο σας απογοητεύτω, δεν έχουν γίνει ολοκληρωμένες συζητήσεις. Ε, ενώ έχει περάσει 1,5 χρόνος μετά από το δημοψήφισμα, έχουν περάσει τόσοι μήνες ανεργοποίηση του άρθρου 50 με εκπλήσει. Βέβαια, του δεν υπάρχει εδώ κανείς βουλευτής υπέρ του Brexit. Ίσως θέλω να το περιμένουμε, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι πάρα πολύ κακό και για τους ε, Βρετανούς, είτε ψήφισανε είτε όχι. Τι γίνεται με την αναγκαία περίοδο υλοποίησης σε σχέση με τον τελικό προορισμό των γιατρών, σε σχέση με την επανεγκατάστασή τους, ε, χρειάζονται κάποιο χρόνο να ε, προγραμματιστούν, ε, γιατί είπατε ότι οι εταιρείες εταιρείες ότι δεν έχει αποκρισταλωθεί το πού θα πάνε. Κύριε Λάφιν, εάν έχουμε no deal, τι θα γίνει με τους ασθενείς, απαντήσεις. Ευχαριστούμε γιατί δεν τόσο την ευκαιρία να επεκταθώ λίγο ε, για την κυρία Μπίρντερ όσον αφορά την έρευνα. Ξεκαθαρίστηκε από τον κλάδο μας το πόσο έχει σημασία η έρευνα, η έρευνα σε όλη την Ευρώπη, πόσο σημαντική είναι. για τις κλινικές δοκιμές, θέλουμε να υλοποιηθούν τα εξαγγελθέντα και η περσμένη εβδομάδα η φαρμακοεποπτεία αυτή η επαγρύπνηση τέλο πάντων ξεκίνησε και αυτό θετικό και προβληματιζόμαστε βέβαια σε σχέση με το Brexit. τι θα γίνει και στους 27 και στο μενό Βασίλειο αν θα συνεχιστεί η συνεργασία. Ως πανεπιστημιακό, έχω συμμετάσχει σε προγράμματα στο παρελθόν. Ξέρω πόσο αξίζουν, ξέρω το πώς ε, συγκεράζεται έτσι η εμπειρία, οι δυνατότητε οι ερευνητικέ. Και ελπίζουμε το θέμα αυτό να φυγεί στις ε, διαπραγματεύσει. Τώρα όσον αφορά το EMA που πήγε στο Άμστερνταμ, είπαμε ότι όχι μόνο η βιομηχανία, αλλά και διάφοροι φορείς πρέπει να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν. Και αυτό αφορά και την προμήθεια των φαρμάκων. Και τώρα τι θα γίνει με το αδίκτυο των ε, κανονιστικών αργών ρυθμιστικών τελικά ε, τελικά η βοήθησε περισσότερο από ότι κάθε υπηρεσία χωριστά ή από το σύνολο και βέβαια η υπηρεσία φαρμάκων της Αγγλίας δεν θα μπορείς να ωφεληθεί πια και είδατε όλοι στις διαφάνειες τι έγινε με τις μεταβιβάσεις αδειών. Είδατε τι έγινε στους 27. Κοιτάξτε τι πρόβλημα θα έχει όταν έρθει η να αντιστραφεί εκείνη η διαδικασία από την ε, δική μας υπηρεσία. Και ακούσαμε τι θα γίνει με τα πρότυπα που θα χειροτερεύσουν. Πρέπει να μας εξασφαλίσει η κυβέρνηση ότι θα νομοθετήσει για να μην πέσουν τα πρότυπα. Μην πέσει το επίπεδο. Να δούμε τι θα απογίνει. Τώρα κάτι τελευταίο, πριν δώσω στον Πολ το λόγο. Ναι, είναι σαφές το θέμα όσο ο κύριος Ντάνς για τη μεταβατική περίοδο. Άμα κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, πώς να προγραμματίσει τη μετεγκατάσταση. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τις ε, εταιρείε, μια που δεν είναι ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο. Άρα, αυτή τη στιγμή το μόνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Βρετανία αποτελεί, θα αποτελεί τρίτη χώρα. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα το συντομότερο. Κύριε Μπίλτερ, πρώτα-πρώτα, όσον αφορά τις επιπτώσεις για την έρευνα. Όσον αφορά τους ε, πανεπιστημιακούς, 16% των πανεπιστημιακών ιατρικών σχολών προέρχονται από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Οπότε, και συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, τελικά είναι θέμα αμοιβαίας αναγνώρισης και ελεύθερης διακίνησης αν δεν μπορούν να διακινηθούν οι άνθρωποι, αν δεν μπορούν να κάνουν την έρευνά τους, δεν θα υπάρξει έρευνα, τόσο απλά. Και στην ε, έρευνά μας ρωτήσαμε τους γιατρούς, τι θα κάνετε μετά τον Brexit, πού θέλετε να πάτε να δουλέψετε. Όχι, δεν ρωτήσαμε μόνο τους ερευνητές, αλλά βέβαια στις ΗΠΑ είναι η πιο μεγάλη αγορά έρευνας. Επομένως τώρα αυτοί που μετακινήθηκαν ήδη θα πρέπει να ξαναμετακινηθούν. Ξέρετε προς τα που άρα ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Τώρα για τον κύριο Τέιλορ και την Ευρωτόμ. Ήλπιζα ότι δεν θα με ρωτήσετε για την Ευρωτόμ γιατί είναι ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα που έχουμε αντιμετωπίσουμε στον Ιατρικό Σύλλογο. Συζήθηκε στην Κάτω αυτό έγινε κάποια ενημέρωση των βουλευτών και εγώ πήγα στην αρμόδια επιτροπή της κάτω βουλής ε, για προφανείς λόγους θα είναι κακό όπως τους είπα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κακό για τους παραγωγούς της Ένωσης γιατί εμείς εισάγουμε πάγο για τη δουλειά μας από Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση παγοκολόνες, τέλος πάντων κάποιο προϊόν πάγου. Και μιλήσαμε σε εκατοντάδε γιατρούς από τότε που αποφασίστηκε το Brexit και κανείς δεν είπε ότι ίσως ωφελήσει το Brexit. Μπορείτε να βγάλετε τα δικά σα συμπεράσματα για το κατά πόσον για τους ασθενείς θα είναι θετικό το Brexit οι επόμενες ερωτήσεις. Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Τα είπα ουσιαστικά όλα ότι ε, δεν έχει να κάνει ε, με το Brexit ή όχι Brexit. Οι Βρετανοί ασθενείς δεν έχουν ε, θετικά πράγματα να περιμένουν έτσι πως είναι τώρα πλέον η κατάσταση. Οι Βρετανοί είναι ε, χρηματοδότης ε, από το Horizon 2020 ε, και βέβαια δεν μιλάμε μόνο για τον ιατρικό τομέα. Αλλά το θέμα είναι εσείς βλέπετε ήδη από τώρα ίσως τις επιπτώσεις της αβεβαιότητας που επικρατεί από τις δύο πλευρές δηλαδή και για τον ακαδημαϊκού κύκλου, αλλά και για τις εταιρικέ ε, ε, σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Ε, υπάρχει κάποια δισταγμό να συμμετέχουν στα προγράμματα, οι κλάδοι. Και στο πλαίσιο της 25ης επαιτίου της Ευρωπαϊκής ε, Καρδιολογικής Εταιρείας μιλήσαμε και με Βρετανούς ε, καρδιολόγους ε, και μας είπαν ότι πολλοί καρδιολόγοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκπαιδευτεί στις χώρες της Πυρωτικής Ευρώπης 25% περίπου, είναι αυτό το ποσοστό. Και τι θα γίνει με τις εμπειρίες που έχουν αποκομίσει. Πάλι υπάρχει εδώ μία ανασφάλεια και τι αβεβαιότητα, τι μπορεί να γίνει ε, με την περίθαλψη ε, μετά το Brexit στις διάφορες ειδικότητε. Και ένα άλλο θέμα σημαντικό δεν είναι μόνο η έγκριση φαρμάκων, η άδεια κυκλοφορία, αλλά τα ακούσαμε και ε, στι τελευταίε παρεμβάσει με τα ραϊδοϊσότοπα και το εμπόριο, μετά το Brexit, πρόσβαση στα, στα φάρμακα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και επίσης ε, με το με το CDC. Τι θα γίνει. Θα υπάρξει ένα παρόμοιο εργαλείο όπως αυτό που έχουμε εμείς τώρα αν υπάρξει περίπτωση ενός σκληρού Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές από τις ε, συζητήσεις ε, για τα, τους οργανισμούς φαρμάκων ε, επικεντρώθηκαν στο πού βρίσκονται. εντάξει, κέρδισε ανικά το χώρο στο Άμστερνταμ, έχασε το Λονδίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως εντάξει, δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχουν συνέπειες και άλλες από αυτό αν δεν αποτελεί, αποτελεί πλαίσιο της δικαιοδοσίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων το Ηνωμένο Βασίλειο στο μέλλον, ποιο είναι το τελευταίο χρονικό όριο κατά το οποίο θεωρείται ότι η σαφήνεια θα ήταν χρήσιμη για να αποφύγουμε την απόλυτη καταστροφή σε σχέση με ε, το καθεστώς, το ρυθμιστικό αλλά και παροχής φαρμάκων για να μην υπάρξουν πάρα πολύ αρνητικές ε, συνέπειες και ενδεχομένως κίνδυνες συνέπειες για τους ασθενείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Μιλήσατε για παράδειγμα ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να επιτύχουμε σε αυτό το επίπεδο ε, ε, ε, ανάπτυξης των φαρμάκων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε. Είπατε ότι δεν προλαβαίνουμε. Ε, είπατε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν ξέρουμε τον προορισμό. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε έναν χάρτη πορείας προς τον προορισμό αυτό. Πόσο όμως θεωρείτε, πόσο, θα θα, πόσο χρόνο θεωρείτε ότι θα χρειάζεται για να υπάρξουν αυτές οι δομές, πόσο προσωπικό θα χρειαστεί για να μπορέσει να υπάρξει ένα σύνολο δομών ε, ε, για να ε, γίνει κάτι τέτοιο. Πόσο το έχετε σκεφτεί αυτό. Κύριε Λάφιν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αρχίσατε την παρουσίασή σας με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και δυνατές ε, ασθένειες ε, σε σχέση με την κατάσταση του NHS ε, στην Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια δεν δημιουργεί ένα πρόβλημα μόνο στο NHS ως προς το πλευρά του, την πλευρά του εργατικού δυναμικού και το Brexit εννοώ. Εγώ πριν έρθω εδώ είδα γενικές, γενικά πόσα προβλήματα πρόσληψης γενικών παθολόγων υπάρχουν και στη δική μου περιφέρεια. Ε, ο Βρετανικός Ιατρικός Σύνογος λοιπόν πώς ιεραρχεί σε τι επίπεδο ιεραρχεί ακριβώς το Brexit ε, ως προς τον τομέα της απασχόλησης είναι ας πούμε το νούμερο ένα πρόβλημα που θα προκύψει. Επίσης, ε, με ενδιαφέρει και η δική σας άποψη ε, ως Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου. Είστε πραγματικά, μπαίνετε και στην πολιτική, την καθημερινή, για, την, ε, για τα ιατρικά προβλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάσταση του ιατρικού τομέα. πώς θεωρείτε ότι η Βρετανική κυβέρνηση έχει αναδείξει το Brexit ως κίνδυνο σε σχέση με την δημόσια υγεία στις διάφορες έρευνες που έγιναν. Θεωρείται, ας πούμε, ε, το Brexit ε, είναι ένας πάρα πολύ ε, επικίνδυνο ζήτημα. Πιστεύω ότι η Βρετανική κυβέρνηση για την ώρα έχει έτσι μια έναν επικίνδυνο εφησυχασμό για το ζήτημα αυτό. αναφερθήκατε στα ευρωπαϊκά δίκτυα ε, αναφοράς. νομίζω 40 νοσοκομεία είναι δικτυωμένα. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ως κέντρο ε, το δίκτυο που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια είναι λοιπόν η ενδεχόμενη απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου αν δεν μπορούμε πια να είμαστε τμήμα αυτού του δικτύου. Από ό,τι κατάλαβα ε, υπάρχουν κάποιες χώρες ΕΟΧ που μπορούν να είναι τμήμα αυτών των δικτύων. Ε, θα χαθεί λοιπόν καινοτομία σε θέματα υγείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αν αυτά τα κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν συμμετέχουν πια σε αυτά τα ευρωπαϊκά δικτύα αναφοράς. Any other questions, Έχετε συνάδελφοι. Αν όχι, να δώσω το λόγο στου προσκεκλημένου μα να μα απαντήσουν. Ευχαριστώ. Για να ξεκινήσω με την κυρία Κάντεμπαχ. Ένα σημαντικό ερώτημα για την έρευνα. Πράγματι, από τις φαρμακοβιομηχανίες σε ό,τι αφορά το IMI για την ε, καινοτόμο έρευνα. Υπάρχει μια σύμπραξη δημοσιοδοτικού τομέα, πολύ μεγάλη επιτυχία, έχει στεφθεί στον τομέα των μελετών και πολλές φορές εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχω έρθει σε επαφή με ακαδημαϊκούς ή επιχειρήσεις που λένε το EMI τι μέλλον θα έχει για αυτούς που είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τις εταιρικές σχέσεις. Γιατί το IMI εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι το κέντρο της εταιρική σχέσης. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο διάλογο πρέπει να συζητηθεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μπορούσε να είναι μια τρίτη χώρα, είναι μια εναλλακτική. Αλλάζει τις δυνατότητες. Δεν θα είναι σε ηγετική θέση το κοινοβούλιο. Το Βασίλειο δεν θα μπορεί να ηγηθεί κανένας προγράμματος, απλά θα συμμετέχει. Είναι μια εναλλακτική, αλλά θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση, ένας διάλογος για τη συμμετοχή στο πλαίσιο εν γέννη. Και ελπίζω η συνεργασία στην έρευνα να μην υποχωρήσει μετά από χρόνια επενδύσεων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δεν έχει αναγνωριστεί αυτό. Τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και η εδραίωση τη συνεργασίας. Πώς θα αντικατασταθούν όλα αυτά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, Πώ θα διαταραχθούν. Αυτό δεν βοηθά την επιστήμη. Να υπάρχουν αυτέ οι ε, τεχνητέ διαχωρήσει σε πολύ παραγωγικέ συνεργασίε ε, και τα δίκτυα αναφορά είναι κάτι που δείχνει ακριβώς την επιτυχία για τις σπανίες ε, παθήσεις, παιδιατρικό ένα ε, θέμα που συζητήθηκε στη Σκοτία. Οι σκοτσέζοι εταίροι έχουν ε, ωφεληθεί πάρα πολύ από το παιδετρικό δίκτυο αναφορά. και αν το χάσω θα είναι πολύ σημαντικέ οι επιπτώσει. και επειδή τα συζητήσαμε εκεί στη Σκωτία εκείνη τη μέρα είδα πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση και σοκ αν σκέφτηκαν ότι αυτά όλα μπορούν να τεθούν ε, σε κίνδυνο Όπω και για το περιβάλλον, όπω και για την ασφάλεια των τροφίμων δεν θα κερδίσει κανεί στην Ευρώπη εάν χάσουμε τη δυνατότητα ανταλλαγή σημαντικών πληροφοριών, δεδομένων ανήγνωση μηνυμάτων, στην φαρμακοεπαγρύπνηση, στον έλεγχο νοσημάτων. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το τραπέζι και ελπίζω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω ποια θα είναι η λύση. Ελπίζω όμως να βρεθεί μια λύση. Αλλιώς υπάρχουν προκλήσεις για όλους. Και αν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πρόγραμμα, τι προβλήματα θα υπάρξουν, αν θα είναι κρίσιμο το ζήτημα. Ουσιαστικά για την FBI η απόφαση αυτή, η μετακίνηση των επενδύσεων δηλαδή, έχει ληφθεί ήδη. Θέλουμε να έχουμε αυτά τα σημεία δοκιμών. Δεν μπορεί μέσα σε ένα μήνα, ούτε και σε μισό χρόνο να γίνει αυτή η μετακατάσταση. Χρειάζεται πολλή χρόνο. Αυτά τα προγραμματίζουμε τουλάχιστον έχοντα ένα ορίζοντα στο μυαλό μας. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες προκλήσεις. Από την έρευνα που έγινε έχουμε προσδιορίσει κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να τις ξέρετε. Ε, προϊόντα δηλαδή τα οποία παρασκευάζονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν δεν μπορούν να εισάγονται στην Ευρώπη, να έρχονται στην Ευρώπη, αυτό θα επηρεάσει σίγουρα τους ασθενείς των 27 χωρών και αντίστροφα. Πρέπει να βρεθεί λύση πραγματιστική, ρεαλιστική. Πόσο χρόνο θα πάρει αυτό όμω θα σας ξαναπώ, εξαρτάται από το πόσο κοντά θα είμαστε. Αν γίνει αυτό που ζητούμε εμείς ως βιομηχανία, δεν θα είναι τεράστιοι σκόπελοι, αλλά αν έχουμε ένα σκληρό Brexit, θα έχουμε να διανύσουμε πολύ ανώμαλο δρόμο. Ευχαριστώ. Για τους καρδιολόγους να απαντήσω. Χρειάζεται 10 χρόνια εκπαίδευση. Αν λοιπόν καρδιολόγοι αποφασίσουν να φύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση αύριο, δεν θα αντικατασταθούν πριν το 2027. Άρα έχει κάποιο ένα καρτελικό πρόβλημα από τώρα μέχρι το 2027, θα μειωθούν πάρα πολύ οι περιπτώσει να μπορέσει να σκεφτεί έναν καρδιολόγο. Αν ήμουν πιο μεγάλο σε ηλικία θα ανησυχούσα τα μάλα. Τώρα δεν έχω κάποιο καρδιακό πρόβλημα, αλλά δεν ξέρω. Για τον κύριο Πάλμερ, για το εργατικό δυναμικό το Brexit αν είναι νούμερο 1, νούμερο 2 ή νούμερο 3 ως κίνδυνος για το εργατικό δυναμικό. Δεν θα έβαζα αριθμούς. Έχουμε θέμα σημαντικό γενικώ με τους γενικούς ιατρούς αλλά και με, τους, ε, με τις ειδικότητε στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Brexit μας αυξάνει τα προβλήματα Διαφορετικά είναι σε κάθε περίπτωση Ιρλανδία, Ουαλία, ε, Σκότη κτλ. Αλλά επιδεινώνονται. Αν δίνετε προτεραιότητα στις ανησυχίες υγείας. Εμείς φροντίζουμε και αυτή είναι η δουλειά μας να το κάνουμε. Εγώ σας είπα. Την επόμενη εβδομάδα συναντήσω έναν υπουργό τη Βετανικής Κυβέρνησης και θα του το, θα τους τα ξαναπώ ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα υγεία στις διαπραγματεύσεις για τον Brexit. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους βουλευτές, ευχαριστώ τα μέλη του πάνελ. Μάθαμε πιο πολλά για την αλληλεξάρτηση μεταξύ μόνο και του Ηνωμένου Βασιλείου και πώς όλοι θα επηρεαστούν. Εάν δεν είναι η ευκταία κατάληξη αυτή του Brexit. Όπως είπα και στην αρχή της συνάντησης. Όλα όσα υπόθηκαν σήμερα, αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες θα τις διαβιβάσουμε στους διαπραγματευτές μας για να αντιληφθούν και αυτοί όπως και εμείς σήμερα πώς έχει πραγματικότητα πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ και πάλι τους ομιλητές και τους βουλευτές. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ίσως. Καλό απόγευμα.